Okay, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, να σας θυμίσω ότι όπως συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται... Ε, τώρα δεν θυμάμαι το ωραίο όνομα που τους έχουν δώσει, έπασε πτώση μεταδίδεται στον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχήν να υιοθετήσουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Εάν όχι, θα χαρούμε πολύ να ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη αυτή. Ευχαριστώ. Έγκριση των πρακτικών. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, ΙΝΙΑΘ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους ε, για την υπομονή τους, γιατί με περίμεναν. για να παρουσιάσω τις πρώτες προτάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους με βοήθησαν για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Είναι πρώτη ανάγνωση, μάλλον έγινε η πρώτη ανάγνωση πριν από τις ευρωεκλογές. Και τότε είχαμε υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση η οποία σε πολλούς ορισμούς είχε καινοτομίες και τώρα που το Συμβούλιο κατέληξε σε ένα συμπέρασμα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία οι απόψεις μας διήστανται και για τα οποία θα πρέπει να βρούμε συνεννόηση. Πρόσφατα βέβαια είχαμε μία πρόσφατη απόφαση του Ευρωδικαστηρίου όπου σε ένα άλλο πακέτο για τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, των, ε, στα αεροπλάνα υπάρχει μία απόφαση η οποία δικαιώνει τη θέση του Κοινοβουλίου που είναι πιο ριζοσπαστική στα θέματα προστασίας των επιβατών. Λοιπόν, βάσει αυτών των δύο στοιχείων θα πρέπει να κοιτάξουμε, να βρούμε μία συνένεση. βασιζόμενοι στις αρχικές μας προτάσεις, αλλά και σε αυτήν την απροσδόκητη βοήθεια που μας δίνει το Ευρωδικαστήριο. Οι διαφορές που έχουμε αφορούν στον εφαρμοστικό τομέα. Εμείς ε, υποβάλαμε μία φιλόδοξη πρόταση για να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όλους τους επιβάτες ε, ε, ορίζοντας ως όριο τους 12 επιβάτες ανά πλοίο, ανά σκάφος. Το Συμβούλιο όμως μας αύξησε τις εξαιρέσεις και ορίζει ως όριο την εφαρμογή της οδηγίας στα σκάφη άνω των 36 επιβατών με πάνω από 3 άτομα πλήρωμα. Υπάρχει και μία εξαίρεση ως προς το βάρος. Πάνω από συγκεκριμένο τον ΑΣ πλοίων. Βέβαια αυτό θα είναι προσωρινό αλλά δημιουργεί σύγχυση στους επιβάτες. Σχετικά με τους ορισμούς, εμείς στο Κοινοβούλιο περάσαμε μία τροπολογία του κυρίου κιρχόπ σχετικά με την ανωτέρα βία, την οποία θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να την δεχθούμε, δηλαδή όταν κόβεται το ρεύμα ή διοικητικό πρόβλημα ή ένα πρόστιμο, ε, ένα άλλο διοικητικό πρόβλημα ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να παρισφρήσει μέσα στα πλαίσια των τεχνικών προβλημάτων υπό το φως αυτής της απόφασης για τα αεροπλάνα θα πρέπει να, τα το ξαναδούμε. Είμαι έτοιμη όμως να ακούσω το τι θα μου πούνε οι συνάδελφοι. Τώρα για το θέμα των αντισταθμίσεων, των αποζημιώσεων, συγγνώμη. Ε, υπάρχει και εδώ ένα θέμα διαφορών, εμείς προστατεύαμε πολύ περισσότερο τα δικαιώματα των επιβατών, ενώ το Συμβούλιο αύξησε την αποζημίωση μέχρι 10 ευρώ. αλλά κατά αυτόν τον τρόπο εξαιρούνται όλες οι τακτικές ε, γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν όλες. Σε περίπτωση ακύρωσης λοιπόν ή καθυστέρησης, η απόφαση του δικαστηρίου βελτιώνει την κατάσταση ε, για τους επιβάτες. Με την απόφαση λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικά διευκολύνει τη δική μας θέση για την προστασία των επίβατων. Τώρα για τα κρουαζερόπλια. Σε αυτή την Επιτροπή εμείς έχουμε και ως αρμοδιότητα την πρόθεση του τουρισμού. Οπότε στα πλαίσια των κρουαζιεροπλίων μπορούμε να έχουμε μια σχετική ευελιξία σχετικά με την βοήθεια, ε, αρρωγή, ενημέρωση. Βέβαια, οι άμεσα αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για όλη αυτή την ιστορία είναι οι ίδιες οι πλειοκτήτριες ε, ε, εταιρείες ε, που οργανώνουν κρουαζιέρες ε, για να βοηθήσουν τους, την πρόσβαση των αναπήρων κλπ. Αλλά και σε αυτά περιμένω να ακούσω τι θα πούνε οι συνάδελφοι. Επίσης, Πρόεδρε, στους συμπληρωματικούς ή προσθετικούς μηχανισμούς προστασίας και διαιτησίας στα δικαιώματα των, πολι... των ε, επιβατών. Σε όλα αυτά λοιπόν, στα οποία, στα οποία εμείς στοχεύουμε ως βουλευτές και ε, που προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών, Ε, για τα θέματα δηλαδή του εφαρμοστικού πεδίου, των αποζημιώσεων, ε, του ορισμού της ανωτέρας βίας και υποποιούς όρους ε, περιορίζεται αυτό το δικαίωμα, θέλουμε να πετύχουμε μία συμφωνία πόσο το δυνατόν περισσότερο να προσεγγίζει τις θέσεις μας. Αυτά Πρόεδρε και περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους ε, τους οποίους ευχαριστώ, ιδιαίτερα την κυρία Βορμανκόλ και την κυρία Μπιλμπάο, ε, που γνωρίζω ότι παρόλο που απουσιάζει λόγω προβλημάτων υγείας, παρακολουθεί τα πράγματα εκ του συνέγγυς. Uh, ευχαριστώ πολύ, Ινιές. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, για να σας ακούσω. Χαίρομαι. που ε, ήρθατε εδώ σήμερα, έχετε, ξεχάσει προσεκτικά, έχετε εξετάσει προσεκτικά τη θέση του Συμβουλίου, που όπως είπατε σε διάφορους τομείς είναι αρκετά διαφορετική από τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει μια συγκεκριμένη αρχή, μεγαλύτερη ευελιξία και για μικρότερα σκάφη και γι' αυτό θέλαμε περισσότερες εξαιρέσεις στο κείμενο. Πρόκειται για μια αρχή την οποία εν μέρη μπορώ να υποστηρίξω. Είναι η αρχή στην οποία βασίστηκε και η τροπολογία μας. Φυσικά θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των επιβατών. Από την άλλη υπάρχουν μικρά σκάφη και θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένη εδώ. Εσείς μιλήσατε για ε, πλοιάρια, ε, για sightseeing κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η λύση μας ε, να ταιριάζει και σε αυτά, διότι αλλιώ κάποιε επιχειρήσει δεν θα μπορούν πια να παρέχουν τι υπηρεσίε του, διότι θα είναι υπερβολικό το διοικητικό άχθος. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε εναλλακτικέ λύσει. και Αυτός είναι ο λόγο για την τροπολογία μα μετά την πρώτη ανάγνωση. Και επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ε, θα μπορέσουμε, πιστεύω, να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, προετοιμάζοντας τη δεύτερη ανάγνωση. Το Συμβούλιο ως κριτήριο έχει οθετήσει το μέγεθος του, του Μιλάνε για 36 επιβάτες, ε, μιλάνε και για τον όγκο του πλοίου, το μέγεθος του πλοίου. Νομίζω ότι κινούμαστε προς την κατεύθυνση με εσά. Ε, τα νούμερα που έχουμε όμως είναι κάπως πιο ε, χαμηλά. Χαίρομαι που αναφέρατε συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά, διότι έτσι μπορούμε να ε, ετοιμαστούμε για τη δεύτερη ανάγνωση, ιδιαίτερα για τα πλοία για sightseeing ή όπου γίνονται οργανωμένες γιορτές. Και τέλος, όσον αφορά τους ορισμούς, η Ευρωπαϊκή τελος οσον αφορα του ορισμου προτείνει ορισμούς ε, ε, έχει εισάγει κάποιους ορισμούς οι οποίοι ε, έχουν τροποποιηθεί και θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν ή από το Συμβούλιο γιατί έχουν γίνει σχετικές τροποποιήσεις στους ορισμούς. Από ό,τι άκουσα εγώ μου φαίνεται ότι θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο της ανασφάλειας δικαίου. Εάν όμως υιοθετήσουμε διαφορετικό όρο για τους ε, οργανωτές ταξιδίων από ό,τι σε άλλες οδηγίες ε, θα έχουμε ανασφάλεια δικαίου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλύτερο να επανέλθουμε στους, αρχικές, στους αρχικούς ορισμούς ε, της Κομισιόν. Θα ήθελα πολύ να ακούσω όμως από την Κομισιόν πώς μπορεί να μας τα εξηγήσει αυτό. Ευχαριστώ κύριο Ελκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γιάλα Σέντερ που είναι η συγγήτρια για την ε, δουλειά της η οποία πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες. Είμαι πεπισμένος ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η έκθεση αυτή. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Είναι αλήθεια ότι στο θέμα αυτό και στο άλλο που θα συζητήσουμε σε λίγο, θα πρέπει να μάθουμε από το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών ε, αερομεταφορών. Δεν ε, Είχαμε σωστές πληροφορίες σχετικά με την ε, υποβολή προσφυγών και έτσι δεν μπορούσαμε να χειριστούμε σωστά το θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μάθουμε από αυτό. Σε μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται ότι η μεγάλη καθυστέρηση ε, ισούται ουσιαστικά με ακύρωση και γι' αυτό δικαιούται αποζημίωση επιβάτης. Ως νομοθέτες θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, έχουν δικαίωμα αποζημίωσης επιβάτες. Μερικές φορές μιλάμε για ε, χρηματική αποζημίωση. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να παράσχουμε ε, βοήθεια, υποστήριξη και ε, ώστε να μπορεί ο τομέας να λύνει τα προβλήματα όταν εμφανίζονται. Και επίσης όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, αρέσει αρκετά η ιδέα του να αφαιρεθούν κάποιες κατηγορίες από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίες ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα μικρά σκάφη. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά τον ορισμό ώστε να μην καταλήξουμε μετά σε μακρές συζητήσεις σχετικά με το αν κάτι επίπτει στο πεδίο εφαρμογή ε, της οδηγίας ή όχι. Να είμαστε λοιπόν απόλυτα σαφείς ε, σχετικά με τους ορισμούς. Θα πρέπει να αναφερόμαστε στον αριθμό των επιβατών, ε, στον όγκο των πλοίων, στο μέγεθος των πλοίων. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό προσεκτικά. Απάντηση δεν έχω. Και δύο τελικές παρατηρήσεις. Αναφερθήκατε σε ένα σύστημα προσφυγών. Ε, εσείς είστε ειδικοί, ίσως ήδη να το έχετε καλύψει, αλλά όπως και να έχει θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα προσφυγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούμε να τις αξιολογήσουμε σωστά, να τις ερμηνεύσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα να τις αντιμετωπίσουμε σωστά. Και δεύτερον, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πάντα ενδιέφερε την ε, Επιτροπή μας, ε, για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα θα πρέπει να φροντίσουμε τα άτομα αυτά, θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεταφορές αυτές υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αυξανόμενο ε, ποσοστό του πληθυσμού. Ο κόσμος γενικά ε, γυράσκει και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την περιορισμένη κινητικότητα. Το ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Θέλετε να μιλήσετε ως και όδηση συγγήτρια? Όχι. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Εύα, θες να μιλήσεις ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις με ενημέρωσαν σχετικά με το περιεχόμενο, συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Δικαιώματα επιβατών και μικρά σκάφη. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Είναι σαφές αυτό σε όλους. Όμως δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την ε, έλλειψη εμποδίων για τους επιβάτες. Θα πρέπει δηλαδή εδώ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εξαίρεση των μικρών πλοιαρίων, ιδιαίτερα εάν είναι τόσο σημαντική η παρέκκληση, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα επιβατών μόνο σε μεγάλα κρουαζιερόπλια. Υπάρχει μια σύμβαση για τα δικαιώματα των ε, ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και άλλων και θα πρέπει να σεβαστούμε τη σύμβαση αυτή. Εάν το Συμβούλιο δεν θέλει να το κάνει αυτό, τότε εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Εγώ δεν το βλέπω τόσο χαλαρά το θέμα ε, ε, να κάνουμε τόσες παρεκκλήσεις ώστε τελικά η οδηγία να ισχύει ε, σε πολύ περιορισμένους τομείς θα ήθελα να καλέσω τους συναδέρφους να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά. Αναφέρομαι σε αυτά συγκεκριμένα στα δικαιώματα αυτών των επιβατών, διότι μου φαίνεται κεντρικό το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε, σε πιθανότατα σε σύγκρουση με το Συμβούλιο, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε υπερβολικό περιορισμό των ε, δικαιωματών αυτών. Ε, θυμάμαι τη συζήτηση ε, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση στα λιμάνια, όλα αυτά ε, συζητήθηκαν Εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ αν εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών ε, δεν υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Ευχαριστώ, Εύα. Η κυρία Έπινγκ. Ε, είσαστε σκιώδης συγητές, συνήθως ε, σε πρώτα σε αυτούς δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα διευκρινήσεις σχετικά με το τι εννοούμε με αποζημίωση. Ακούσαμε επανειλημμένα τη λέξη αυτή. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Τι σημαίνει όμως την πράξη. Σημαίνει ότι επιστρέφεται το συνολικό ποσό ότι προσφέρεται στον επιβάτη η εναλλακτική λύση. Ή για παράδειγμα φτάνει κανείς ε, με πλοίο και δεν μπορεί να ε, δεν προλαβαίνει το αεροπλάνο του. Ε, τι γίνεται. Θα πρέπει ο καταναλωτής να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για την αποζημίωση αυτή. και επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφισημία ως προς τον όρο ακύρωση. Εάν δεν είναι σαφές αυτό στους πολίτες, στους καταναλωτές, Οι καταναλωτέ μπορεί να ετοιμάζονται για ένα ταξίδι, τελευταία στιγμή να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτό δεν είναι μόνο απογοήτευση αυτή η καθεαυτία, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο τι είδους αποζημίωση μπορεί να λάβει. Εγώ έχω ταξιδιέψει πολύ, ε, επανειλημμένα χρειάστηκε να ακυρώσω τις ε, μετακινήσεις μου και πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να ε, λάβει κανείς την αποζημίωση την οποία δικαιούται σύμφωνα με τον νόμο. Ας καταλήξουμε λοιπόν ε, σε έναν καλό ορισμό. Ευχαριστώ κύριος Βαντάλεν. Να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγητριά η οποία εστίασε την προσοχή της στην ουσία του προβλήματος, για την οποία θέλω να μιλήσω και εγώ. Τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το θέμα. Γι' αυτό μπορώ να βεβαιώσω ότι η συγκεκριά όντως εστίασε την προσοχή της στην ουσία του πράγματος. Χρειάζεται προσοχή εδώ. Να μην προκύψει σύγχυση μεταξύ εσωτερικών θαλασσιών οδών και θαλασσίων μεταφορών. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, να σκεφτόμαστε τα 36 άτομα, τους 300 τόνους κλπ. Διότι υπάρχουν μικρές θαλάσσιες, ε, με με εσωτερικές λατινές οδοί που εξυπηρετούνται μόνο από μικρά σκάφη, αλλά υπάρχουν και νερά τα οποία είναι πιο επικίνδυνα. Ε, τα νερά είναι πιο επικίνδυνα πόσο σχέλνεται στο Βέλγιο. Έχουμε νερά ταραγμένα στα οποία χρειαζόμαστε τουλάχιστον 300 τόνους για να μπορέσει κανείς να κυκλοφορήσει με ασφάλεια. Κακώς λοιπόν δεν έχει προκριθεί η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών εσωτερικών υδατινών οδών. Τώρα, όσον αφορά τι αποζημιώσει, φυσικά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Χρήζει περαιτέρω εξαίρεση. Το θέμα για είναι το εξή. Όταν υπάρχει καθυστέρηση, ο σκοπός είναι να καλυφθεί η καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωσή μας, σε διαστολή με τα αεροδρόμια, όπου όταν ένα αεροπλάνο χάσει την χρονοθυρίδα του, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αποζημίωση εδώ. Πιστεύω ότι στην περίπτωσή μα, όταν πρόκειται για καθυστερήσει, μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και πολλέ φορέ μικρέ καθυστερήσει μπορούν να αντισταθμιστούν. Αυτά προ το παρόν και ευχαριστώ. Κύριε Φώστερ. Πρόεδρε, εντάχει, καταρχήν συμφωνώ με τον κύριο Βαντάλεν όσον την διάκριση των σκαφών για τα ανοιχτά ύδατα από αυτά για τις για την οδούς. Εδώ δυστυχώς βλέπω ότι έχουμε αντιγράψει ουσιαστικά τα κείμενα για τις τα μεταφορές. Είναι σαν να έχει γίνει αντιγραφή σε ορισμένα σημεία. Υπάρχουν τώρα περιπτώσεις όπως η κακοκαιρία, ορισμένε κυριακέ συνθήκε για τι οποίε πρέπει να χωρίσουμε εξαιρέσει. Ω προ το Συμβούλιο τώρα, δεν είναι σαφή η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι μάλλον τα πράγματα. Γιατί εμεί έχουμε στο μυαλό μα φυσικά τι δυσμενεί κυριακέ συνθήκε, αλλά ε, τι γίνεται με την περίπτωση απεργία ή τρομοκρατική απειλή. Μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα. Δεν αναφέρονται αυτά παρά το γεγονό ότι είναι προφανή Δεν θέλουμε λοιπόν οι επιβάτες να μην παίρνουν αποσμίωση λόγω του ότι ήταν ασαφή η διατύπωσή μας εδώ. Τώρα όσον αφορά το μέγεθο του πλοίου, τη χωρητικότητα του πλοίου και το πλήρωμα, ε, εξαρτάται περί τίνο πρόκειται. Και να με βοηθήσει κάποιος από, από γιατί δεν ήμουν εδώ την περασμένη φορά. από πού βγήκε το 500 μέτρα ε, για τον ορισμό του πολύ σύντομου ταξιδιού. Είναι το πλάτος ενός ποταμού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι και το σωστό. Δεν έχω αντιπρόταση. Απλώ αναρωτιέμαι πώ καταλήξαμε σε αυτό το 500 μέτρα. Δεν ξέρω αν πήγε κανεί μετροτενία και... ή θα πάρει μετροτενία για να δει αν ήταν 500 501 τα μέτρα. Λίγο παράξενο μου φαίνεται αυτό το 500. Εν πάση περιπτώσει, τέλο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι οι επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα. Πολλοί από εμάς έχουν ταξιδέψει με κρουζιρόπλια μεταξύ άλλων. Ε, ο λόγος για τον οποίο άνθρωποι με αναπηρίες πηγαίνουν τέτοιες ε, κρουαζιέρες ακριβώς επειδή υπάρχει περιποίηση και επειδή ακριβώ ε, υπάρχει συγκεκριμένη ειδική προσπάθεια για να διευκολυνθούν αυτοί οι επιβάτε με περιορισμένη κινητικότητα να λάβουν μέρο σε τέτοιου είδου ε, κρουαζιέρε σε ε, ποτάμια ή αλλού. Πρόεδρο. Εγώ προσωπικώ συμφωνώ με την ισχύτρια όσον αφορά την ανάγκη ευελιξία, ειδικά εναντί της, του τομέα τη κρουαζιέρα. Περιμένουμε και από αυτού μάλιστα, προτάσει πρέπει να σα πω. Χρειάζεται πάντω προσοχή, όσον αφορά τον τομέα αυτόν συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, ε, για να μην προκύψει ένα κείμενο ιδιαίτερα δεσμευτικό, με πρόσχημα τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, για παράδειγμα. Λοιπόν, να το δούμε. Τώρα για το 500 δεν έχω ιδέα. Είναι αυτό το οποίο έφερε η κυρία Φώστερ. Αλλά πιστεύω ότι τώρα πια Υπάρχει τεχνολογία, δεν χρειάζεται κανεί να πάρει με το ταινία, να κολυμπήσει, να διασχίσει ένα ποτάμι. Υπάρχουν ε, ειδικέ συσκευέ με τι οποίε με το πάτε μια σκανδάλη ε, μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια μέτρου αν είναι 500-590 μέτρα. Δεν είναι όμω αυτό το θέμα. Σε περιφέρειες όπως το Μέρσι, σε εξαιρούνται οι μεταφορές από τη μία οχθή στην άλλη σε εκβολές ποταμών, για παράδειγμα. Όπως ήταν προηγουμένως. Να το δούμε αυτό. Γιατί εκεί έχουμε εξαιρέσει. Τώρα, ε, από την Κομισιόν, κύριε Διαχούντο, κύριε ο λόγος σε εσάς. Έχουμε μαζέψει πολλές ερωτήσεις για εσάς, περισσότερες από ό,τι για την εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Euh, euh, euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επανέλθω σε όλη αυτή την ιστορία της πρότασης εντάσσεται στο πολιτικό πλαίσιο ε, της Κομισιόν που είναι πάντα υπέρ των επιβατών, ευθυγραμμίζεται με την ανακοίνωση του 2005 για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών. Αυτές οι δύο προτάσεις του Δεκεμβρίου 2008 για τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, των ε, πλοίων, η άλλη πρόταση για τους επιβάτες των αεροπλάνων και, για τις και των οδικών μεταφορών δεν ήταν ε, εύκολο να διατυπωθούν. Γιατί Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τη Σουηδική Προεδρία, η οποία σε λίγους μήνες κατάφερε να διαμορφώσει μία συνένεση γύρω από αυτό το ντοσχέ, εν ώψη μίας ε, οριστικής λύσης. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι ένας, αποτελεί μεγάλη πρόοδο για όλο τον τοσχέ. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή, τον κύριο Τεσενέ, που σε πρώτη ανάγνωση κατάφερε να συσπυρώσει το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Απριλίου γύρω από αυτές τις προτάσεις. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, η συγγήτρια, έκανε μια εξαιρετική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολιτικής συμφωνίας. Το κείμενο του Οκτωβρίου από το Συμβούλιο είναι ένα κείμενο το οποίο απομακρύνεται από το κείμενο που πρότεινε η Κομισιόν και υποστήριξε το Κοινοβούλιο. Αυτό αφορά και το εφαρμοστικό πεδίο, όπως εξάλλου υπόθηκε, και τις ε, καθυστερήσεις ε, λόγω καιρικών συνθήκων, αυτό το έβαλε το Συμβούλιο, και το θέμα των αποζημίσεων. Επίσης και το θέμα των κατοφλίων, των ορίων για αποζημίωση. Εμείς δεν διαφωνούμε ότι υπάρχει μία διαφορά μεγεθών στο κείμενο που, διαπραγματευτήκαμε, που διαπραγματευόμαστε. Πρέπει λοιπόν εμείς να καταφέρουμε να βρούμε το 2010 μία συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων. Θεωρούμε ότι οι διαφορές δεν είναι τέτοιες που θα διακυδεύσουν την τελική συμφωνία ή θα την καθυστερήσουν υπερβολικά. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μία συμφωνία αρκετά σύντομα και για να επανέλθουμε σε μερικές λεπτομέρειες που εύστοχα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Είναι φανερό ότι η Κομισιόν στους ορισμούς προσπαθεί να προσαρμοστεί με ορισμούς που έχουν διατυπωθεί σε άλλα κοινοτικά κείμενα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μία ε, συμβατότητα με την οδηγία 90 314 για τα οργανωμένα ταξίδια. Το Συμβούλιο επίσης ε, συμμερίζεται αυτήν την άποψη και θελήσαμε να αξιοποιήσουμε και την όλη εμπειρία που έχουμε στην προστασία των ε, επιβατών ε, των αερογραμμών. Και ένα τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε, που αφορά στα 500 μέτρα και στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Κατά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, τα 500 μέτρα ελήφθησαν υπόψη για να καλυφθούν και οι διάδρομοι εσωτερικής ναυσιπλοείας, όπως επίσης και οι μικρές διαδρομές, τόσο δηλαδή οι θαλάσσιες ε, μεταφορές όσο και οι ποτάμιες. Για να καλυφθούν λοιπόν τα σύντομα ταξίδια, οι σύντομες ε, διαδρομές, ε, μπήκε αυτό το κριτήριο των 500 μέτρων. Αυτά προς στιγμή. Ε, κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέλφους για τα χρήσιμα σχόλια. Και θέλω να τονίσω εκείνες τις ε, πλευρές που είναι και οι πιο σημαντικές ε, για τους πολίτες. Εμείς ε, ελπίζουμε να μακροημερεύσουμε ούτω ώστε όταν θα γίνουμε κι εμείς άτομα με περιορισμένη κινητικότητα να μπορέσουμε να καρποθούμε των μέτρων που θα αποφασίσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και σας ευχαριστώ και για την αισιόδοξη τοποθέτησή σας. Διότι εγώ όταν διάβαζα παράλληλα τα κείμενα, ε, έβλεπα πολύ μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αυτών που αποφασίσαμε εμείς στην πρώτη ανάγνωση και του κειμένου του Συμβουλίου. Και όχι μόνο δηλαδή στις ε, ε, θαλάσσιες μεταφορές αλλά και στις αεροπορικές μεταφορές και οδικές μεταφορές. Φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος Καντσάν μετά θα το, το, θα το σχολιάσει το θέμα, αλλά καλό είναι το Κοινοβούλιο να θέσει αυτές τις προτάσεις ως πακέτο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις ε, δυσκολίες. Και όταν φτάσουμε πια ε, στην εξέταση των τροπολογιών να μιλήσουμε ε, σαφώς με το Συμβούλιο και να ακολουθήσουμε τη γραμμή του πακέτου για την προάσπιση των τροπολογιών έναντι του Συμβουλίου. Ένα λοιπόν συνολικό πακέτο για την προστασία των επιβατών. Θα έρθω σε επαφή ε, σύντομα και με τους κοιόδης εισηγητές ε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία για τα δικαιώματα των επιβατών που πάντοτε υπερασπιστήκαμε αλλά και στην ανάγκη να παραμείνει και ζωντανός αυτός ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός στα θέματα, στον τομέα της ναυσιπλοείας. Πράγμα το οποίο το έχουμε παλέψει και στο παρελθόν, δηλαδή με προγράμματα όπως ο Μαρκοπόλο. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους. Θα ήθελα όμως να έχουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερους ορισμούς για να αποφύγουμε την νομική ανασφάλεια, όπως είπε και ο συνάδελφος Χαδράουι. Υπάρχει επίσης ε, και το θέμα της υποβολής παραπώνων που και αυτό εκκρεμεί και θα θέλαμε να το διαπραγματευτούμε. Εγώ θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους και θα καταθέσω τις απαραίτητες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κανσιόν για τα δικαιώματα των Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω συμφωνώντας ε, με την κυρία ε, Γιάλα σχετικά δηλαδή με την προσέγγιση πακέτο. Πρόκειται για την τέταρτη ρύθμιση σχετικά με τα τρένα και τα αεροπλάνα και τα πλοία που συζητιούνται τώρα. Αλλά για τα λεωφορεία, ενώ το Συμβούλιο για τις άλλες προτάσεις έχει καταλήξει σε μια πολιτική συμφωνία, για τα λεωφορεία δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα στοιχείο ότι θα μπορούσε να προκύψει συμφωνία στις 17 Δεκεμβρίου. Εμείς ξεκινάμε από το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης της 23 Απριλίου όπου μόνο 30 άτομα καταψήφισαν την έκθεση του συναδέλφου Αλμπερτίνη τότε. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτήν τη βάση θα πρέπει να παραμείνουμε και να συνεχίσουμε. Ζητώ λοιπόν από σήμερα επίσημα την εντολή από την ε, Επιτροπή για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ανάγνωση. Εγώ είχα δύο άτυπες συναντήσεις με την Σουηδική Προεδρία και είχα και επαφή θέσα και με τον αρμόδιο της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Τα βασικά ζητήματα που συζητιούνται αφορούν στο εφαρμοστικό πεδίο και κυρίως αφορούν στο καθεστώς ευθύνης. Χρειάζεται λοιπόν να ορίσουμε τι είναι η περιφερειακή, με τι είναι οι περιφερειακές μεταφορές, γιατί ενώ για τις αστικές μεταφορές ε, υπάρχει μία αρκετά σαφής, ε, ένας αρκετά σαφής ορισμός για τις ε, διαπεριφερειακές επικοινωνίες ε, δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια μία διαφορά μεταξύ των αστικών ε, και υπεραστικών μεταφορών ε, και των περιφερειακών μεταφορών. Αλλά όμως εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω το 75% των μεταφορών. Δεν είναι σωστό να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι θα πρέπει να καταλήξουμε Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διαχωρίσουμε εμείς τις μεταφορές και να αφήσουμε τη διακριτική ευχέρεια των κρατών την δυνατότητα να επηρεάσουν ε, με την κατάσταση, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει και το δικαίωμα προς των επιβατών ε, που θα λαμβάνεται υπόψη, διότι εμείς ε, πρέπει να προστατεύσουμε τους επιβάτες και όχι τα λεωφορεία ή τις εταιρείες. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά, τη γνώμη μου θα πρέπει να, τα, να πάρουμε όλες αυτές τις μεταφορές, τους τρόπους μεταφοράς υπόψη μας. Για την ευθύνη, την αντικειμενική ευθύνη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την προστασία του χρήστη. Να προστατεύσουμε λοιπόν έλεγα τους επιβάτες και, από, και σε περίπτωση δυστυχημάτων αλλά και σε περίπτωση απώλειας ε, των αποσκευών. Υπάρχει ήδη νομοθεσία για τα οχήματα, αλλά υπάρχουν και δύο παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και που είναι σημαντικές. Και που αφορούν στην, στον ορισμό ενός συγκεκριμένου ποσού σε περίπτωση δυστυχήματος με βαριές επιπτώσεις, όπως επίσης και η άμεση βοήθεια που θα πρέπει να διασφαλίζεται. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το αντικειμενικό κριτήριο και αυτή, αυτά τα δύο κριτήρια, δηλαδή προστασία των προσώπων από τη μια και των αποσκευών από την άλλη. Επίσης προστασία των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Μιλάμε για 127 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 50 ε, εκατομμύρια είναι ανάπηροι. Και όλοι αυτοί θα αυξηθούν αν λάβουμε υπόψη και τη γύρανση του πληθυσμού. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτω ώστε τα λεωφορεία να είναι προσβάσιμα από όλα τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Αν μέσα από την προσέγγιση πακέτο με την έκθεση της ε, κυρίας Αγιάλα για την αυσυκλογία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα και για την Ολομέλεια. Περιμένουμε εμείς τον ορισμό και από την πλευρά του Συμβουλίου, διότι το Συμβούλιο ακόμη δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ελπίζουμε να συμφωνήσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. για να προχωρήσουμε τις δύο εκθέσεις μαζί. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινή θέση και για τους δύο κανονισμούς. Η γενική φιλοσοφία, κατά τη γνώμη μου, επειδή μιλούμε για δικαιώματα των πολιτών, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ως επίκεντρο τον πολίτη επιβάτη. Και είναι πολύ σημαντικό όλοι οι συνάδελφοι, κυρίως οι σκιώδεις συζητητές, να στείλουν τις παρατηρήσεις τους, ούτω ώστε να έχουμε συμφωνήσει ε, πριν από, την, ε, από αποφαση, την απόφαση του Συμβουλίου. Κυρία Σαρατσάνη. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως έλεγε και ο κύριος Καντσάν, τα βασικά προβλήματα είναι ποιος έχει την αντικειμενική ευθύνη και το εφαρμοστικό πεδίο. Το Συμβούλιο θέλει το διαχωρισμό μεταξύ των περιφερειακών και των διαπεριφερειακών συγγνώμη, ε, μεταφορών και των αστικών και περαστικών συγκοινωνιών. Χρειάζεται να έχουμε λοιπόν μία μελέτη για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διευρύνουμε το πεδίο του κανονισμού. Τώρα η Σουηδική Προεδρία θέλει ε, να υποχρεώσει αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες να αποζημιώνει με 120.000 ευρώ ε, αναεπιβάτη σε περίπτωση θανάτου. Θέλουμε επίσης ε, να γίνει μία διάκριση ε, από τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Οπότε το Συμβούλιο θέλει να κάνει κάθε κράτος μία ταξινόμηση των περιφερειακών ε, συγκοινωνιών στην ε, κάθε χώρα, δηλαδή αριθμός στάσεων, χιλιόμετρα κλπ. Τους δύο κανονισμούς τους παρουσίασε μαζί η Κομισιόν, αλλά για τα λεωφορεία καθυστέρησε το Συμβούλιο. Ελπίζουμε στις 17 Δεκεμβρίου να αποφασίσει και για τις μεταφορές με λεωφορεία. Επειδή τώρα το Κοινοβούλιο θέλει να συζητήσει τα δύο ντοσιέ παράλληλα, εγώ συμφωνώ στο να συζητηθούν σε πακέτο τα δύο μέτρα, γιατί αυτό θα το καταλάβουν και καλύτερα ήδη οι πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Meissner. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι όλοι περιμένουμε το Συμβούλιο να καταλήξει οριστική θέση, ε, η οποία θα αποτελέσει την προϋπόθεση για την συνέχεια των εργασιών μας. Ε, στην πρώτη ανάγνωση πράγματι υπήρχε ε, μεγάλη συνένεση και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εξέταση του θέματος αυτού των δικαιωμάτων των επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν. Θα ήθελα να αναφέρω πολύ σύντομα ότι στον ορισμό θα πρέπει να φαίνεται σαφώς ποιος είναι υπεύθυνο για θέματα ευθύνης, ποιος είναι υπεύθυνο για τις μεταφορές, σε ποιον, σε ποιον θα πρέπει να στρέφονται δηλαδή οι επιβάτες. Επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί το τι γίνεται σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων κλπ. Θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς ορισμούς. Επίση από τη συζήτηση προέκυψε ότι είναι αποφασιστική σημασίας αυτό που θα συζητήσουμε κατά τη δεύτερη ανάγνωση να είναι πραγματοποιήσιμο, να είναι ρεαλιστικό, να ε, είναι αυτό που θέλουμε τελικά, να είναι εφαρμόσιμο. Στις αερομεταφορές είναι κάπως λιγότερο δύσκολο σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ακυρώσεων να ε, βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος μεταφοράς. Ε, εδώ πέρα δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Θα πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε να προβλέπουμε σωστές λύσεις στην οδηγία. Επίσης, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, κάποιοι θέλουν να αφαιρθούν οι αστικές και προαστικές μεταφορές. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, επιβατών, ε, σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Ήδη πολλοί άνθρωποι έχουν ε, τέτοιους περιορισμούς λόγω της δημογραφικής αλλαγής. Θα έχουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών και στις θελάσσιες μεταφορές και στις μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία. Ε, υπάρχει και το θέμα, για παράδειγμα, των μητέρων, με, ε, ε, των ανθρώπων με παιδικά καροτσάκια. Είναι σημαντικό να αποφελούνται όλοι από τις μεταφορές. Όσον αφορά την ε, κοινή συζήτηση και για τις θαλάσσιες μεταφορές ε, θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Φυσικά θα απλοποιηθεί έτσι η κατάσταση για τους ε, ασφαλιστές, για τους οργανωτές ταξιδιών. Τότε θα πρέπει να εξετάσουμε εάν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε διαφορετικούς κανόνες για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τις μεταφορές με πούλμαν. Ε, φυσικά είναι πάντα καλύτερο να έχει κανείς ε, ενιαίου κανόνε, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, αν είναι δυνατόν αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Φυσικά περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα παρουσιάσει το Συμβούλιο. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα καλό πακέτο το οποίο να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα σε αυτό το θέμα είναι η δυσκολία να γίνει διάκριση ανάμεσα στις περιφερειακές μεταφορές, ε, αστικές ε, μεταφορές και τις ε, μεταφορές σε μεγάλων αποστάσεων με πούλμαν. Διότι σε πολλές περιφέρειες υπάρχουν ενώσεις μεταφορών που ε, ασχολούνται με όλες τις μεταφορές αυτές, που καλύπτουν όλες τις μεταφορές αυτές. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, εάν ε, για μια διαδρομή χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μέσα, δύο διαφορετικά πούλμαν και μιλάμε για δύο διαφορετικά είδη μεταφορών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα υπάρχοντα δικαιώματα των επιβατών για να βρούμε μια καλή λύση η οποία να αποτελέσει βήμα πρόοδου. Διότι μπορούμε να συναντήσουμε σημαντικές δυσκολίες σε πολλές περιφέρειες. Έχουμε μεγάλες ε, ενώσεις μεταφορών που καλύπτουν ε, και μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων και αστικές. μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι δύσκολο για τους επιβάτες να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα αυτό ως προς την υπερασπίση των δικαιωμάτων. Τίθεται λοιπόν το θέμα ποιο είναι υπεύθυνο και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνεται ο επιβάτης. Δεύτερο θέμα που μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, που ήδη αναφέρθηκε στο, στα πλαίσια των θαλασσίων μεταφορών, είναι η ευελιξία. Η ευελιξία έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι, για παράδειγμα, στην Ελβετία, στους σιδηροδρόμους, η ευελιξία έχει εφαρμοστεί με πολύ θετικό τρόπο. Οι επιβάτες μπορούν μόνοι τους να επιλέξουν. Θέλουν ως αποζημίωση ένα γεύμα, έναν καφέ, ένα γλυκό μέχρι το επόμενο τρένο. Θέλουν ε, χρηματική αποζημίωση, επιστροφή ή θέλουν βοήθεια για να προλάβουν κάποιο άλλο τρένο. Εδώ η ευελιξία είναι πολύ θετική. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και εις βάρος των επιβατών, εάν το ένα είδος αποζημίωσης είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί, ενώ το άλλο είναι πολύ εύκολο. Μπορεί λοιπόν ε, ο επιβάτης να προτιμάει ένα και στο χέρι παρά και καρτέρι σε μερικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, είναι δύσκολο καν να βρω το γραφείο στο οποίο θα πρέπει να ε, προσφύγω. Γι' αυτό ίσως είναι πολύ πιο εύκολο απλά να δεχτώ την προσφορά να πάρω το επόμενο λεωφορείο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρίες μας από τους σιδηροδρόμους και τις αερομεταφορές. Θα πρέπει να φροντίσουμε η ευελιξία να είναι προς όφελος του επιβάτη και όχι να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν παραθυράκια ως προς ε, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όπως ήδη είπα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό είναι σημαντική πρόκληση για το μέλλον και ε, και εγώ ίδια ε, ε επαφελούμε, διότι όταν ε, ταξιδεύω με βαριές βαλίτσες, πάντα χαίρομαι για τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί για αναπήρους, διότι έτσι η μετακίνησή μου με μια βαλίτσα, με ένα παιδί, είναι πολύ πιο εύκολη. Υπάρχει η φιλανθρωπική διάσταση, αλλά Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ε, ορισμό των ε, μεταφορών στο μέλλον. Οι μεταφορές στο μέλλον θα πρέπει να περιλαμβάνουν ε, το στοιχείο της πληροφόρησης, ενημέρωση για τους προορισμούς, για τους, για τους δρόμους κλπ. να φροντίσουμε να είναι οι μεταφορές εύχριστες για τους επιβάτες. Προσπαθήσαμε αυτό στην πρώτη ανάγνωση να το διευκρινίσουμε, αλλά το σημείο αυτό ε, εκρεμεί ακόμα και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη σχετικά με αυτό που θα δούμε από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπράτπορν. <clears throat> Πρόεδρε, σαν τα έχω ξανακούσει κάπου όλα αυτά. Τα επιχειρήματα τα ξανακούσουμε όταν μιλούσαμε για θεωροπορικές μεταφορές, για τα τρένα, τι αποζημιώσει και τώρα ξαφνικά τα ίδια με τα λεωφορεία, τα πούλμαν κλπ. Δεν έχω αντίρρηση επί της αρχής, βεβαίως. Οι επιβάτε πρέπει να αποζημιώνονται όταν κάτι πάει στραβά με το ταξίδι τους. Όμως όλα αυτά έχουν και κάποια πρακτική πτυχή. Πώς εφαρμόζονται λοιπόν στην πράξη πώς ξεκινούμε, πώς κατεβαίνουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο στο τοπικό. Να σκεφτούμε λίγο πώς λειτουργούν τα πούλμαν και τα λεωφορεία. Όταν συζητούσαμε τους σιδηροδρόμους, αν θυμάστε, είχα επικρίνει και τον εισηγητή, τον κύριο Στέρξ, την εποχή, όταν είχε έρθει κουβέντα στα τοπικά σιδηροδρομικά ταξίδια, τις ε, μικρές διαδρομές, γιατί προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε τα πάντα ακόμα και για αυτέ τι απλέ τοπικέ διαδρομέ. Και το ίδιο κάνουμε δυστυχώ και εδώ με τα πούλμαν και τα λεωφορεία. Εγώ θα πρότεινα να περιοριστούμε στα διεθνή ταξίδια. Ή τελειώ πρέπει να δημιουργήσουμε διαφορετικέ κατηγορίε όσον αφορά την ενημέρωση, τι ρυθμίσει, τι αποζημιώσει. Θα πρέπει και εδώ δηλαδή για τα και τα πούλμαν, να ρυθμίσουμε ένα σωρό ατελείωτες λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να κατέβουμε σε τοπικό επίπεδο και να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τα πάντα. Το τι θα γίνει, η αποζημίωση θα ζητήσει κάποιος όταν αγοράζει ένα στήριο που κάνει ένα δυο ευρώ ή τρία. Ο κ. Λίχτεμπεργκερ μίλησε για τα σχετικά στην Ελβετία, αλλά και εμεί από το Λονδίνο στο Δημβουργό έχουμε λεωφορεία τα οποία χρεώνουν 5 λίρε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να υποχρεώσουμε μια εταιρεία να πληρώσει ξενοδοχείο και διατροφή για ένα εισιτήριο που κάνει 5 λίρε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Χρειάζεται κατά περίπτωση αντιμετώπιση. Ε, εννοείται φυσικά ότι Κάποια πράγματα πρέπει να προβλέψουμε σχετικά με τις αποζημιώσεις. Να υπερμηνθούμε εννοείται των δικαιωμάτων των επιβατών, αλλά όχι με τρόπο ισοπεδρικό. Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, ξέρετε στον Ηνωμένο Βασίλειο, ε, έχουμε ψήφιση ρύθμιση, χάρη στην οποία οι άνω των 65 μπορούν να ταξιδεύουν δωρεάν λίγο πολύ παντού. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Κάποιος ο οποίος ταξιδεύει δωρεάν ανά την επικράτεια θα αποζημιώνεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν ο οποίος έχει πληρώσει ένα μεγάλο ποσό για την ίδια διαδρομή. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για την εφαρμογή. Δεν με απασχολεί η αρχή, με την οποία συμφωνώ, αλλά μακριά από ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Ανησυχώ κύριε Πρόεδρε. Όχι για την αρχή, το ξαναλέω αλλά ακούω να βαβαριζόμαστε με προτάσεις από την Κομισιόν, οι οποίες αποτελούν δάνειο, αντιγραφή από προηγούμενες διατάξεις, από ένα άλλο χώρο. Προσπαθούμε λοιπόν με ένα ράβε ξύλο να τις προσαρμόσουμε εδώ με τρόπο μη πρακτικό. Είναι τελέσφορη προσπάθεια να προδιαγράψουμε όλες τις ρυθμίσεις για διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης, διαδρομών και υπηρεσιών, επίπεδα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναπηρίες και δεν μιλάμε μόνο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, μιλάμε για ανθρώπους που δεν ε, βλέπουν ε, ή που ε, δεν ακούν, των οποίων η κινητικότητα είναι περιορισμένη ή που έχουν διανοητική αναπηρία. Εγώ είχα την αίσθηση ότι τα έχω ξαναδεί αυτά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μιλήσαμε για τις αερομεταφορές και για τα δικαιώματα των επιβατών στον τομέα αυτών. Συμφωνούσαν όλοι τότε ότι οι ορισμοί δεν είναι σαφείς και εδώ βλέπω το ίδιο πρόβλημα. στις σημερινές παρεμβάσεις, αλλά και στο σχέδιο έκθεσης ε, βλέπουμε ότι αναφέρονται τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Αλλά αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι σε σχέση με την πρώτη ανάγνωση βλέπω ότι πολλές προτάσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη, παρότι το Κοινοβούλιο έχει οθετήσει τις προτάσεις αυτές. Επιμένω Οι άνθρωποι με αναπηρίες και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο να δουν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Στην δεύτερη ανάγνωση τέτοια δικαιώματα εφαρμόζονται μόνο στις ε, μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Τι γίνεται όμως με τις αστικές και περιφερειακές μεταφορές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν πολύ συχνά τις μεταφορές αυτές. Και το τρίτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω και που θα ήθελα να, όπου θα ήθελα να παρουσιάσω και γραπτώ σε μία πρόταση είναι τα άρθρα 18 και 19 που αναφέρονται σε όλους τους τομείς. Το άρθρο 10 λέει ότι, ε, ότι η ελευθερία ε, κινητικότητας είναι μια από τις εμελιώδεις ε, ελευθερίες των ανθρώπων. Δεύτερον, άρθρο 18... Αναφέρεται εδώ η κατάρτιση το, του προσωπικού. Ακόμα και αν ε, ένα λεωφορείο ε, έχει ε, προβλεφθεί για άτομα με περιορισμένη κινητικο... με αναπηρίες, εάν ο οδηγός δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά, εάν το προσωπικό δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, τότε οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αυτή. Και η τρίτη ε, πτυχή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα είναι ότι όταν ε, γίνονται ατυχήματα, θα πρέπει να προβλέπουμε κάτι. Για παράδειγμα, εάν κάποιο σε ένα πυρικό καροτσάκι ε, τραυματιστεί ή κάτι τέτοιο, ε, θα πρέπει να λαμβάνει σχετική αποζημίωση. Τα θέματα αυτά όμως δεν αναφέρονται στο σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Και εγώ συμφωνώ ότι καταρχήν συνδέονται άμεσα αυτά τα δύο ντοσιά, αλλά να σας ε, θυμίσω ότι η κατάσταση διαφέρει διότι στην Ισπανία υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο και στη χώρα μου, αλλά όπως και στη Γερμανία πολλές φορές, τα άτομα με περιορισμένες ε, κινητικές ε, ε, δυνατότητες προτιμούν αυτή την οδική μεταφορά που είναι μεταφορά από πόρτα σε πόρτα. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα όχι μόνο των ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε γενικά την κινητικότητα και τις ίδιες πληροφόρησης, ώστε όλοι να ενημερώνονται, θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή και την Κομισιόν σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται αυτή η βαθμιαία εφαρμογή. τα στη χώρα μου τα λεωφορεία τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν λιγότερο ή μικρότερο εισόδημα αλλά που έχουν και προβλήματα κινητικότητας. Επίσης σε απομακρυσμένα χωριά ε, ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι όλο αυτό το δίκτυο λεωφορείων. Θέλω να ξέρω λοιπόν σε ποιο βαθμό γίνεται και μία διαβάθμιση Ε, ευελιξία της επιχειρήσεις, φυσικά διασφαλίζοντας βέβαια τους επιβάτες, αλλά μία σιγουριά για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα τόσο η Κομισιόν όσο και ο εισηγητής να εξετάσουν την ιδιομορφία αυτή αυτού του τύπου μεταφοράς που είναι εντελώς διαφορετική ως προς την τυπολογία του χρήστη. Υπάρχει και η στενή επαφή επίσης μεταξύ οδηγού και επιβατών που δεν έχουμε σε κανένα άλλο μέσος μεταφοράς. Ja, ο κύριος Κράμερ. Ναι, μου κάνει εντύπωση που δεν ε, εποφελούμαστε περισσότερο από τις ε, εμπειρίες μας. υιοθετήσαμε την απόφαση για ε, τις ε, σιδηροδρομικές ε, μεταφορές. Υπάρχουν εκεί κάποια θετικά και αρνητικά ζητήματα. Καταφέραμε να ισχύουν κάποια πράγματα για το σύνολο των μεταφορών Αλλά για παράδειγμα, παίρνει κανείς ε, το τρένο από το Βερολίνο στις ε, Βρυξέλλες, ε, λαμβάνει αποζημίωση από τις Βρυξέλλες μέχρι το Άχεν, από το Άχεν όμως μέχρι τη Λιέγη όχι, από τη Λιέγη μέχρι τις Βρυξέλλε πάλι ναι. Και πάλι εδώ μιλάμε για διεθνείς μεταφορές. Στις μικρές χώρες το 90% είναι διεθνείς μεταφορές, ενώ στις μεγάλες χώρες είναι μόνο το 10%. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε από την αρχή όλη τη συζήτηση. Δεύτερον, ε, τα κέντρα διατησία. Στη, στις μεταφορέ μεταφορές ε, έχουμε κάτι τέτοιο, οι αερομεταφορέ όμω αρνούνται να έχουν κάτι τέτοιο. Τρίτον, για τι συνδρομικέ μεταφορέ θα πρέπει μέχρι το τέλο τη χρονιά να εφαρμοστούν τα δικαιώματα των ε, επιβατών για κάποιες ε, χώρες ε, μπορεί να δοθεί κάποια παρέκκληση. Αλλά εγώ άκουσα ότι ακόμα δεν υπάρχει διεθνής ε, πληροφόρησης παρότι, πληροφόρησης παρότι όλα είχαν αποφασιστεί. Λοιπόν, όταν μιλάμε για χρήματα, δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε οικονομικά τις επιχειρήσεις, θέλουμε να, οι μεταφορές να γίνονται στην ώρα της. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορούν να παραπονεθούν ότι ε, πρέπει να πληρώσουν ε, αποζημίωση. Μέχρι τώρα μέχρι Τώρα ε, κάνω τη δουλειά του εις βάρος των ε, επιβατών. Ε, στο Βερολίνο λένε για παράδειγμα ότι αν, φύγει υπερβολικά νωρί το λεωφορείο, αν δηλαδή εγώ φτάσω 10 η ώρα και έχει ήδη φύγει το, λεωφορείο που ήταν προγραμματισμένο στι 10, εγώ μπορώ να πάρω ταξί. Την πρώτη φορά να το πληρώσει επιχείρηση, την δεύτερη θα ζητήσει από τον οδηγό να το, να το πληρώσει. Δεν ε, υπάρχει δικαιολογία ότι ήταν το τελευταίο μου δρομολόγιο και ήθελα να γυρίσω νωρί στο σπίτι. Όσον αφορά την ε, περιορισμένη κινητικότητα, το 30% των ε, επιβατών στις δημόσιες μεταφορές έχουν κινητικό περιορισμό. Και δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους σε καροτσάκι, μιλάμε για ηλικιωμένους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κυλιόμενες σκάλες, τις μητέρε με παιδιά, καροτσάκια. Χρειάζεται πολλής χρόνο και πολύ υπομονή Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι μιλάμε για το 30% και ο αριθμό αυτός αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε πολύ αυστηροί. Και εδώ θα ήθελα να φέρω το παράδειγμα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουν τι εμπειρίες του από το Βιετνάμ. Κάθε λεωφορείο κάθε λεωφορείο ε, έχει προδιαγραφέ για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και όχι για του αναπήρου, όχι για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, αλλά για τους βετεράνους. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Πρόεδρε, είπαμε στην αρχή η Ευρωπαϊκή το Ευρωπαϊκό το Συμβούλιο μάλλον, με συγχωρείτε, έστειλε έκθεση πρόοδου. Βέβαια, δεν έχουμε οριστική εικόνα, αλλά ορισμένοι βουλευτές σχολήσαν το θέμα του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογή αυτού του κειμένου, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μιλάμε για πούλμαν και λεωφορεία. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει και το θέμα της επικουρικότητας. Αφορά τις περισσότερες διαδρομές. Λοιπόν, με την ευκαιρία να σχολιάσω τα εξή. Το πρώτο αφορά τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα. Ακούστηκαν αξιόλογα σχόλια και όντως υπάρχουν τέτοιοι επιβάτε με διαφορετικού περιορισμού, αλλά ο κ. Λίχτενμπέργκερ θυμάμαι ότι είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι με βαριά προβλήματα, οι οποίοι θα χρειάζονταν ε, ειδικού τύπου οχήματα, βιοταχή κλπ. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδε χιλιάδες επιβατών με μικρότερα προβλήματα και φυσικά αν ε, ένα αναπηρικό μαξίδιο χαλάσει υπό τι ζημιέ. Πρέπει ε, να αποσμιωθεί ο ενδιαφερόμενο. Αλλά ποια είναι η ευθύνη τελικά του οδηγού. Είναι εκπαιδευμένο ε, να βοηθάει στην επιβίβαση και υποβίβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Στις αεροπορικέ μεταφορέ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, ξέρετε. Διότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και έχουν βαριά προβλήματα κινητικότητας έχουν κάποιον μαζί τους συνήθως. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι ένας οδηγός λεωφορείου δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά νοσηλευτής ή ειδικό σε θέματα μεταφοράς ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν άτομα, να το πω αλλιώ, που χρειάζονται βοήθεια από ξεχωριστά άτομα και ο οδηγό δεν είναι πάντοτε σε θέση να το κάνει. Ύστερα, το θέμα της ευθύνης και της ασφάλισης για την εν λόγω ευθύνη που πρέπει να συστήσουν οι εταιρείε. Χρειάζεται πολύ προσοχή για το τι ουσιαστική ευθύνη αναλαμβάνουν. Άκουσα μάλιστα τρομακτικά νούμερα για απώλεια αποσκευών. Άκουσα κάποιο ανατετόριο 1.300 ή 1.800 ευρώ. Η διαφορά, προσέξτε όμως, είναι ότι εδώ αντιγράφουμε και πάλι τον αεροπορικό τομέα στον οποίο 99,9% των ανθρώπων έχουν ασφάλιση αποσκευών. Εδώ πέρα όμω κανεί δεν το κάνει στα λεωφορεία και τα πούλμαν. Ποιο λοιπόν φέρει την ευθύνη αν γίνει κάποιο ατύχημα, αν χαθεί μια αποσκευή βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των αερομεταφορών και των πούλμαν και των λεωφορείων, διότι α, για ιστορικού λόγους εξελίχθηκαν τελείω διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το ανώτερο το οποίο θα προκρινεί το Συμβούλιο, γιατί δεν ξέρω πού βρίσκεται το, το Συμβούλιο, ποια είναι η του. Αυτά προς το παρόν. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ακούσω την άποψη τη Κομισιόν. Παρακαλώ, κύριε Ζήκε. Με δύο λόγια. δράτω τις ευκαιρίες της συγκεκριμένη συζήτηση για να κάνω μια πρόταση. Ξέρετε, είτε πρόκειται για αερομεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, πούλμαν ή λεωφορεία θαλάσσιες μεταφορές, όλοι συμφωνούμε επί της γενικής αρχής. Συμφωνούμε δηλαδή η λεωφορεια θελασσιες μεταφορες ολοι συμφωνουμε επι της γενικης αρχης συμφωνουμε δηλαδη η έλλειψη διακρίσεων, η εξυπηρέτηση των ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητα, τα θέματα των καθυστερήσεων, ακυρώσεων, ατυχημάτων, απόλυση πρόσφυγων κλπ. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει χρειάζεται ενημέρωση και βεβαίω ισχύουν οι αρχέ που διαπούν τα δικαιώματα των επιβατών. Από την άλλη πλευρά, το πεδίο εφαρμογή πρέπει να εξειδικευθεί ανάλογα με τον τύπο της μεταφοράς και το ίδιο ισχύει και με τις αποζημιώσεις. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε καλύτερα το ζήτημα και ευχαριστώ τον συνεργαστή εκ των προτέρων, διότι όπως είπα, το πεδίο εφαρμογή και το αντικείμενο των αποσμιώσεων, το περιεχόμενο και το ύψο των αποσμιώσεων, πρέπει να προσαρμοστεί στον τύπο τη υπηρεσία που συζητούμε. Εμείς τακτοποιήσαμε τους σιδηροδρόμους, τις αερομεταφορές. Είμαστε τώρα στις χερσαίες μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Καλό θα ήταν λοιπόν να διατυπώσουμε ενδεχομένω έναν γενικό χάρτη δικαιωμάτων των ταξιδιωτών, των επιβατών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, θα στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη έχει πολιτική για τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί είναι κάτι το οποίο διαχέεται στην ομίχλη των νομοθετημάτων μας. Να θυμίσω λοιπόν ότι υπάρχουν δικαιώματα των επιβατών. Και το ξαναλέω διότι οι σχετικές πληροφορίες, η ενημέρωση, χάνεται από εδώ και από εκεί, είναι κατακρεματισμένη και δεν είναι αποτελεσματική. Εμείς θέλουμε να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες μας. Γιατί, για να λειτουργεί η δημοκρατία ως προς και τα δικαιώματα των επιβατών. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με σχετικά απλό τρόπο θα έλεγα θα μας επέτρεπε να συγκεντρώσουμε, να ενερμονίσουμε το θέμα του χειρισμού των καταγγελιών και των παραπώνων. Έστω λοιπόν και εκ των υστέρων, αφού καταρτήσουμε όλους αυτούς τους σχετικούς κανονισμούς, να αποφασίσουμε να καταρτήσουμε ένα γενικό χάρτη που θα προβλέπει δικαιώματα και αποζημιώσεις και για τους τέσσερις τομείς μεταφορών. Θα μας βοηθούσε να είμαστε πιο σαφείς εναντί των πολιτών μας και θα μας έκανε και πιο ορατούς ο πολιτικής απόψεως εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριο Σαπίν. Πρόεδρε, Κύριε Κραμα. είπε αυτό που ήθελα ακριβώς με ναι, πόσο αφορά τις ΗΠΑ. Υπάρχει σύνδεση και εδώ μεταξύ προφανώς πεδίου εφαρμογή και προσβασιμότητας για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Και ο Σκράμερ μίλησε για τις ΗΠΑ, στις οποίες έζησα λίγο πριν εκλεγώ εδώ. Στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, όλα τα λεωφορεία έχουν ειδικέ ε, εξέδρες ε, Ανεψουμένε πλατφόρμες για την επιβέση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Και αυτό δεν είναι μόνο για αυτούς, αλλά και για ορισμένους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν τα ίδια, ίσως και μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχουν δυο πλατφόρμες που τους μεταφέρουν από το πεζοδρόμιο στο λεωφορείο. Και κανείς δεν ε, παραπονιέται για την καθυστέρηση ότι δεν δουλεύει το ένα ή το άλλο. Θεωρείται όλα αυτά και κοινωνικό, με συγχωρείτε, και εκτιμένο, απολύτως κανονικά και καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεκαθαρίσουμε το αντικείμενο αυτού του κανονισμού, τι σημαίνει τοπικό, τι σημαίνει περιφερειακό. Περιφερειακό σημαίνει και διαπεριφερειακό από την μία επαρχία στην άλλη δεχομένω. Φυσικά στην Ολλανδία είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι από τη Γαλλία και Γερμανία, αλλά να τα δούμε όλα αυτά παρακαλώ. Επίσης, πρέπει να αφήσουμε να ισχύσει σε κάποιο βαθμό και η επικουρικότητα. Αφού δούμε φυσικά πώς θα λειτουργήσει αυτός ο κανονισμός στην πράξη. Είναι βέβαιο ότι είναι αδύνατον ένα πλαίσιο με ένα νομοθέτημα να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν ευελιξία. Ιδιαίτερα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, ναι, 10 δευτερόλεπτα για ένα σύντομο ερώτημα. Αν συμπεριλάβουμε τα λεωφορεία που παίρνουν τα σύνορα, αυτό σημαίνει ότι για Μάλτα, Κύπρο, Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία το κείμενο αυτό δεν θα ισχύει επειδή δεν έχουν ακριβώ λεωφορεία τα οποία ε, από τη μια χώρα στην άλλη. Υπάρχουν ε, κάποια λεωφορεία που παίρνουν τα σύνορα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγα είναι, αλλά υπάρχουν. Ε. η κυρία Χάπμαν. κυρια η λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε με αυτή την πρόταση εμείς θέλουμε να συμπληρώσουμε όλα, ε, σε όλα τα μέσα μεταφοράς τα δικαιώματα των επιβατών. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ίση μεταχείριση μεταξύ των ε, ε, μεταξύ των επιχειρήσεων και των επιβατών πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν να διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το πεδίο. Για το θέμα της ευθύνης των πρακτορείων λεωφορείων σε περίπτωση τραυματισμών ή απώλειας αποσκευών. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές μέσα στην Ένωση <coughs> και αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα στους ε, επιβάτες, κυρίως στις διεθνείς μεταφορές και είναι ένα ουσιαστικό σημείο της πρότασής μας. Σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τις ουσιαστικές γραμμές της πρότασης και το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι και η Κομισιόν μάλλον θεωρεί ότι η πρώτη σειρά τροπολογιών είναι πολύ σημαντική για τα δικαιώματα των επιβατών. Και ήταν δύσκολη η συζήτηση, τουλάχιστον για την πρώτη σειρά των μέτρων, αλλά θέλω να ευχαριστήσω του Ειδική Προεδρία που πραγμα... παραδειγματικά προχωράει στην αναζήτηση ενός συμβιβασμού και για να ξεκαθαρίσω μερικές παρεξηγήσεις. Η πρόταση σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει αποζημιώσεις, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τον καταβλισμό σε ξενοδοχείο. Θέλουμε να έχουμε εμεί έναν ενιαίο νόμο που να εφαρμίζεται παντού. Ελπίζουμε το Συμβούλιο να καταλήξει στις 17 ε, Δεκεμβρίου σε μια πολιτική συμφωνία για να μπορέσετε να αποφασίσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη δεύτερη ανάγνωση βάσει των δύο προτάσεων και η συνέχεια για μας θα ήταν να καταλήξουμε το 2010 στην οριστική αποδοχή του κανονισμού <coughs> βελγική προεδρία. Όλες αυτές οι προτάσεις χρειάζονται ένα συμβιοβιστικό πνεύμα από όλου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία και η Κομισιόν θα εκφράσει και αυτή το δικό της το πνεύμα και σίγουρα θα διευκολύνει στην εξέβρεση συμφωνίας. Έγινε ερώτηση σχετικά με το πακέτο. Η Κομισιόν είναι πολύ ευήκοη σε αυτό. Πιστεύουμε εμείς ότι σε μερικές μέρες για την πρόταση για τα λεωφορεία θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Δηλαδή θα δούμε επίσης εάν το μπλοκάρισμα των λεωφορείων θα αποτελέσει τροχοπέδι για την πρόθεση της ε, ναυσιπλοείας. Και για να απαντήσω στον κύριο Κράμερ, μέχρι την Πέμπτη θα δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τον κανονισμό Μπράι και την εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη και για να απαντήσω και στην πρόταση του κυρίου Ρικέ πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αποδείξει ότι η Ευρώπη τελικά ε, υπολογίζει στα δικαιώματα των επιβατών και του χρόνου θα έχουμε και μία μεγάλη καμπάνια πληροφόρησης ε, για όλα τα μέσα μεταφορών ε, που θα προβάλλει τα δικαιώματα των επιβατών. Συνάδελφοι, καταρχήν, ένα λεπτό θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Νομίζω θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την κυρία Αιάλα Σέντερ Κυρία Χάπμα, μπορείτε παρακαλώ να κλείσετε το μικροφωνό σας. Ευχαριστώ. Ε, απλά βλέπω την ωραία σας εικόνα εδώ μπροστά μου, στις οθόνες. Θα ήθελα να δώσω στους, ε, στην και στους σκιώδεις εισηγητές να διαπραγματευτούν. Αν συμφωνείτε μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Επίσης θα ήθελα αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε τα δύο σε ένα πακέτο αυτή τη στιγμή και εάν υπάρχει κοινή θέση και για τα δύο να διαβαστούν και τα δύο μαζί, όχι ξεχωριστά. Ακούω τι λέει η Κομισιόν Ε, ότι μπλοκάρισμα στα λεωφορεία μπορεί να ε, καθυστερήσει αδικαιολόγητα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά ναι, η ζωή είναι δύσκολη στο Συμβούλιο. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε τα θέματα αυτά ως πακέτο και να επιτρέψουμε στου, στο, στους εισηγητές και στους σκιώδεις εισηγητές να προχωρήσουν με τη βάση αυτή. Αν συμφωνείτε, ε, να προχωρήσουμε έτσι. Ε, ο κύριος Κάνση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε για αυτή τη διευκρίνηση που θεωρώ απαραίτητη, ε, θεωρώ απόλυτα σωστή, διότι το να αφήσουμε στη μέση του δρόμου τα λεωφορεία και να προχωρήσουμε με τα άλλα μέσα μεταφοράς δεν είναι σωστό. Εμείς τα λεωφορεία θέλουμε να κολλήσουμε με τους υπόλοιπους κανονισμούς. Ελπίζω λοιπόν, θεωρώ μάλλον ότι η συζήτηση σήμερα ήταν πολύ χρήσιμη, σημαντική και για μένα, αλλά θέλω να τονίσω ότι εμείς δεν αναζητούμε να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα κάποιους για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των επιβατών. Απλώς θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευθύνες, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες όσοι ασκούν αυτού του ίδιου στις δραστηριότητες, διότι πολλές φορές το κάνουν πραγματικά με ελαφρομυαλιά. Τώρα σίγουρα είναι σαφές ότι όποιος ε, σφάλει πληρώνει. Τα πάντα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς ε, θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις πλευρές του ζητήματος για να υπερασπιστούμε ε, τα, τους πάντες, κυρίως αυτούς που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Εμείς δεν θα μπούμε εδώ ούτε στην αρχιτεκτονική των πόλεων, ούτε στη μηχανική των λεωφορείων. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε ορισμένα δικαιώματα να παραμείνουν ε, ε, εγγυμένα και να διασφαλίνονται στο μέλλον. Αστικές και περαστικές συγκοινωνίες, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας κανονισμούς ήδη υπάρχοντες ε, που προστατεύουν τα δικαιώματα των αναπήρων. Ε, αν δεν αφομοιώσουμε λοιπόν αυτούς τους παλιούς κανονισμούς δεν χρειάζεται καν να το εξετάσουμε το θέμα. Φυσικά και θα πρέπει να το διαχωρίσουμε στα δύο, να το εξετάσουμε χωριστά αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε λίγο και τον ορισμό της περιφερειακής συγκοινωνίας. Καταλαβαίνω τον διεθνή, τις, διεθνείς συγκοινωνίες, καταλαβαίνω αστικές, υπεραστικές συγκοινωνίες. Το περιφερειακό πρέπει να αλλάξουμε. Διεπόμενος από αυτό το πνεύμα και ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι 557 ψήφοι υπερψήφισαν αυτή την έκθεση και το άρθρο που περιλαμβάνει το άρθρο 2 όπου λέγεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να βγάλουν από το καπέλο της οδηγίας τις ε, αστικές και περαστικές ε, μεταφορές. Εμείς αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε. Το αν πληρώνεις εσύ δύο στερλίνες ένα εισιτήριο δεν σημαίνει ότι άμα σκοτωθείς δεν θα πρέπει να σε αποζημιώσουν. Ευχαριστώ κύριε Καντσάν πολύ έγκυρο το επιχείρημά σας. Ε, χρήσιμο που μας ενημερώνετε, που μας θυμίζετε τι ψηφίσαμε τελικά, διότι μερικές φορές παρασύρεται κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνήσαμε ότι οι συγητές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τους κοιόδες συγητές και συμφωνήσαμε ότι προς το παρόν θα διατηρήσουμε τα δύο αυτά ως πακέτο. Το επόμενο θέμα είναι ε, τα, ε, τα τέν ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πακέ. Νομίζω ότι είναι εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχουμε λιγότερο από μία ώρα, διότι ε, έχουμε στις 5.30 τη συνεδρίαση των συντονιστών. Να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώρα, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε επί μία ώρα. Εάν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και λιγότερο και θαύματα συμβαίνουν παρακαλώ, αν αποχωρείτε, αποχωρήστε ήσυχα και τι συζητήσει σας έξω, όχι μέσα στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σπακέ. try... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συμβάλλω στη δημιουργία του θαύματο με μια σύντομη παρουσίαση λιγότερο από 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση αυτή, το αποτέλεσμα της ε, πρόσκληση υποβολής ε, προσφορών 2009 για το TNT πρόγραμμα και το πολιετές πρόγραμμα. Ε, έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε δύο εντύπα τα οποία δίνουν μια επισκόπηση της διαδικασίας αυτής και αναφέρονται και τα προγράμματα τα οποία διατηρούνται για χρηματοδότηση, αναφέρεται και ποια προγράμματα υποβλήθηκαν τα οποία όμως δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Η παρουσίαση αυτή γίνεται από το 2007 που συμφωνήθηκε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει την παρουσίαση αυτή. Πρωτού πάμε σε ε, διαδικασία επιτροπολογία. Ε, Στι 7 Δεκεμβρίου θα πάμε λοιπόν στην Επιτροπή Οικονομική Βοήθεια, όπου ελπίζουμε να έχουμε την ε, υποστήριξη των 100 μελών για τη χρηματοδότηση και κατόπιν θα ξεκινήσει η διαδικασία τη επιτροπολογία. Τρία προγράμματα είχαμε το 2009. Το ένα ήδη υιοθετήθηκε και μάλιστα ε, με επιμέρους αποφάσεις για τη χρηματοδότηση έχουν ήδη ληφθεί. 500 εκατομμύρια ευρώ συμφωνήθηκε να δοθούν από την Κομισιόν σε σχετικά, ε, ε, σε σχετικά έργα. Αυτό 1η Ιουλίου παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο. Ο προϋπολογισμός ε, λοιπόν TNT συμβάλλει στην δημιουργία έργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι συμβάλλει και στην έξοδο από την οικονομική κρίση. τα δύο επομένω προγράμματα είναι κάπως μικρότερα. Έχουμε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 80 εκατομμύρια και έχουμε τη δόση του 2009 του πολιετούς προγράμματος σε τρία στοιχεία ε, οδικές μεταφορές, ε, έξυπνες ε, μεταφορές ε, και η διαχείριση της κυκλοφορίας με IATRS. Να σας αναφέρω σύντομα την διαδικασία. Η επιλογή φέτος ήταν πολύ δύσκολη για το πολιτές πρόγραμμα. Είχαμε 80 εκατομμύρια στη διάθεσή μας με βάση το πρόγραμμα εργασίας που υιοθετήθηκε στην αρχή του 2009 στην Επιτροπολογία με τα κράτη-μέλη και με εσάς. 96 προτάσεις είχαμε που ζητούσαν χρηματοδότηση 359 ε, εκατομμυρίων ευρώ, 80 ε, εκατομμύρια όμως ήταν ε, διαθέσιμα. Κάναμε λοιπόν την συνήθεια αξιολόγηση σε δύο στάδια που κάνουμε. Καταρχήν εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τα επιμέρους προγράμματα με βάση τα κριτήρια του κανονισμού TNT. Η εξωτερική αυτή αξιολόγηση επέτρεψε να κατέβουμε από, τα 90, από τις 96 προτάσεις σε 59 προτάσεις για χρηματοδότηση που είχαν υποβληθεί. Οι 59 αυτές προτάσεις ε, αντιπρόσωπευαν ακόμα τα 246 εκατομμύρια ευρώ και πάλι ήμασταν λοιπόν πολύ πάνω από τα 80 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα ε, με την υποστήριξη της ε, εκτελεστικής υπηρεσίας TNT ε, καταφέραμε από τα 59 αυτά έργα να επιλέξουμε 32 προτάσεις. Στο έντυπο που σας ανέφερα έχετε ένα πρώτο κατάλογο των έργων αυτών μαζί με το ποσό της χρηματοδότησης που προτείνεται και θα βλέπετε και κάποιες παρατηρήσεις που εξηγούν γιατί διατηρήθηκαν τα προγράμματα αυτά. Και τα 32 αυτά προγράμματα είχαν προταθεί από την ε, εξωτερική αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκαν με την εσωτερική διαδικασία της Επιτροπής ε, από το προσωπικό της DG Trend και της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον. Βλέπετε και το κατάλογο των ε, έργων που απορρίφθηκαν είτε γιατί απορρίφθηκαν από την, κατά την εξωτερική αξιολόγηση, είτε επειδή απορρίφθηκαν ε, από την Επιτροπή για διάφορους λόγους. Καταρχήν, προσπαθήσαμε να ε, ακολουθήσουμε πολύ στενά τις ε, προτεραιότητες ε, πολιτικής και τους στόχους ε, που έχουν ήδη καθιερωθεί. Δεύτερον, κάποια από τα έργα φάνηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα στον τομέα του παρεμβάλλοντος. Ε, απορρίφθηκαν λοιπόν και έπρεπε τελικά να, και, να κάνουμε και κάποιες επιλογές για λόγους προϋπολογισμού. Ήταν λοιπόν δύσκολη η δουλειά μας, πολλά προγράμματα, πολλές ανάγκες στα κράτη-μέλη. Ε, θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποιες στατιστικές σχετικά με το τι είδους προγράμματα χρηματοδοτούμε. Σε μεγάλο βαθμό φέτος ε, θα αφοσιωθούμε στις μελέτες. Το 72 τα 100 των 80 εκατομμυρίων ε, θα δοθεί σε μελέτες. Υπάρχει το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης όπου αναφέρονται πολλοί μελέτης οι μελέτες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν επικεντρώνονται περισσότερο σε μελέτες που ε, ετοιμάζουν το έδαφος και πολύ συχνά είναι πολύ χρήσιμες για να επιταχύνουν την προκατακτική φάση έργων που ε, τελικά πραγματοποιούνται. Έχουμε λοιπόν 22% ε, προγραμμάτων που είναι έργα και μετά έχουμε ένα μικρό αριθμό που περιλαμβάνουν και μελέτες και έργα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις μεταφορές που είναι ενδιαφέρον τομέας. Θα δείτε ότι έχουμε προτάσεις για όλους του, για όλους τους τρόπους ε, μετακινήσεων, ιδιαίτερα ε, επικεντρωνόμαστε στις οδικές μεταφορές και τους σιδηροδρόμους. Ε, αν δείτε τι προτάθηκε και τι διατηρήθηκε, θα δείτε ότι είχαμε αρκετά προγράμματα που αφορούσαν τα αεροδρόμια. Δυστυχώς μόνο ένα διατηρήθηκε ε, πέσαμε λοιπόν από το 3% στο 1,6% διαχείριση αερομεταφορών και εδώ μπορέσαμε να διατηρήσουμε μόνο ένα. Εσωτερικά ύδατα, αυτό, ε, εδώ είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία. Είχαμε 7 προτάσει από τι οποίε διατηρήθηκαν οι 5, συνδυασμένες μεταφορές 8 προτάσει από τι οποίε διατηρήθηκαν οι 3, ε, λιμάνια είχαμε 8, διατηρήθηκαν 3, Σιδηρόδρομοι διατηρήθηκαν 11 Ε, προγράμματα. Ε, βλέπουμε όμως ότι το σύνολο ότι το συνολικό μερίδιο τελικά ήταν 53% στις ε, προτάσεις που διατηρήθηκαν. Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον. Αυτά είναι γενικά τα στοιχεία του, του ετησίου προγράμματος. Δεν θα, Δεν θα αναφερθώ στα επιμέρους προγράμματα. Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο και τις σχετικές παρατηρήσεις. Φυσικά μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, αργότερα. Να αναφερθώ τώρα στο πολυετές πρόγραμμα, το οποίο ήταν το δεύτερο πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Έχουμε τρεις ε, τομείς, ε, ITS, οδικές μεταφορές ε, και ε, διαχείριση των μετακινήσεων. θαλάσσιες μεταφορές. Εδώ δεν καταφέραμε να αποφορήσουμε τον προϋπολογισμό. Έξι προτάσεις είχαμε, μόνο μία προτάθηκε για χρηματοδότηση από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ο λόγος ήταν ότι για τα άλλα προγράμματα η συμμετοχή των κρατών μελών δεν ήταν η απαραίτητη ή δεν ήταν γεωγραφικά ισορροπημένες οι προτάσεις ή δεν ευθυγραμμίζονταν με το, την ε, έννοια αυτών των θαλασσίων μεταφορών. Μπορέσαμε λοιπόν να διατηρήσουμε πρόγραμμα μόνο για 17 εκατομμύρια από τα 30 εκατομμύρια που είχαμε αρχικά. Αυτό είναι λυπηρό αποτέλεσμα και στην Κομισιόν εργαζόμαστε πάνω στο πρόγραμμα του, της επόμενης ε, χρονιάς. Ε, θα πρέπει τώρα να αφιερώσουμε χρόνο ώστε να μάθουμε από τα αποτελέσματα αυτά, ώστε να διασφαλίσουμε πέρσι η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά το ITS είχαμε τρεις προτάσεις. Η μία προτάθηκε για χρηματοδότηση, πρόκειται για τη δεύτερη φάση του Easy Way που χρηματοδοτήθηκε ήδη το 2007. Έχει ολοκληρωθεί τώρα και με την ε, πρόσκληση αυτή υποβολή προτάσεων μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Σημειώνω ότι πριν επιβεβαιώσουμε τα 100 εκατομμύρια για την δεύτερη φάση θα ε, πραγματοποιήσουμε μία μελέτη ε, για την πρώτη φάση για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο και να διασφαλίσουμε τα ενιαία πρότυπα ITS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο πρόγραμμα, ε, ERTS ε, ακολουθεί ε, μία πρώτη πρόσκληση η αποβολή προτάσεων που έγινε το 2007. 260 εκατομμύρια είχαμε τότε και εδώ πέρα Είχαμε 52 ε, προτάσεις για 367 εκατομμύρια ευρώ, 240 εκατομμύρια ήταν ε, διαθέσιμα. Καταφέραμε λοιπόν να περιορίσουμε τον αριθμό ώστε να παραμείνουμε εδώ του προπολογισμού. Μετά τη σημερινή παρουσίαση και τις ε, παρατηρήσεις σας θα περάσουμε στην Επιτροπή Οικονομικής Αρρωγής στις 5 Δεκεμβρίου και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσουν τις προτάσεις αυτές κατόπιν το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα και ελπίζουμε η Επιτροπή να μπορέσει να υιοθετήσει τις σχετικές αποφάσεις τον Ιανουάριο, κάτι που θα επιτρέψει στις επιμέρους αποφάσεις να ληφθούν από την εκτελεστική υπηρεσία ε, TNT για να υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα να μιλήσω για να ενημερώσω την Επιτροπή σας σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του 2010 που παρουσιάστηκε πέρσι στην ε, Επιτροπή Οικονομικής Αρρωγής. Ε, τώρα έχουν περάσει προτάσεις αυτές ε, στην Επιτροπολογία, μπορεί να τις έχετε δει ήδη. Βρίσκονται, έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Δύο προγράμματα προτείνουμε το 2010 αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι πολιετές, το οποίο θα καλύπτει σύστημα πληροφόρησης για τα εσωτερικά ύδατα, για τα για τα ποτάμια και έχουμε και το δεύτερο μισό για τα airspace blocks, ε, όπου προτείνονται 20 εκατομμύρια για τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και επίσης έχουμε ένα ετήσιο πρόγραμμα για το 2010, το οποίο είναι κάπως ιδιαίτερο με την έννοια ότι καλύπτει δύο πολύ συγκεκριμένα οικονομικά μέσα. Το το IGTT μέσω εγγυήσεων, το οποίο εφαρμόζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, ήδη διαθέσαμε 105 εκατομμύρια στην ε, τράπεζα. Ε, είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμή και έχουν ζητήσει 50 εκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότησης που θα διατεθούν στα πλαίσια αυτού του ετησίου προγράμματος. και, και εδώ έχουμε μια νέα εξέλιξη, θα συμβάλλουμε από τον προϋπολογισμό TEN-T με 80 εκατομμύρια στο Ταμείο Μάργκεριτ, το ταμείο που προτείνεται στο ε, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης. και η FW της ε, Γερμανίας, ε, το, ο αντίστοιχος φορέας ε, στη Γαλλία και υπάρχουν και πολλοί άλλοι χορηγοί από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πολωνία, την Ιταλία κλπ. Αυτό είναι πάση είναι το Ταμείο Μαργκερίτ. Η Κομισιόν προτείνει να, να συνεισφέρουμε με 80 εκατομμύρια στο Ταμείο αυτό. Αυτό προκύπτει, προβλέπεται στον κανονισμό TNT το 1% των 80 εκατομμύρια, το 10% τους ε, ε, ε, είναι 80.000, 3,5% είναι η μόχλευση Ε, καταλήγουμε με, μετά από όλου του υπολογισμούς σε 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ προγράμματα. Προβλέπετε λοιπόν το 1,5% του προϋπολογισμού για το Ταμείο Μαργκαρίτ. Ήθελα να το αναφέρω αυτό σήμερα, ώστε να μην ε, περάσει απαρατήρητο αυτό από την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ υποψήφιοι ομιλητέ. Για το ετήσιο πρόγραμμα τα πράγματα δεν θα είναι και πολύ εύκολα. Βαδίζουμε σε ανώμαλο έδαφος για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εικόνα. Να ακούσουμε όμως τι έχουν να πούν οι βουλευτές, κύριε Κρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τις 5.30. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις πληροφορίες. Πολύ σύντομα. Το αποτέλεσμα της επιλογής ήταν περίπου αυτό που περιμέναμε, ιδιαίτερα όσον αφορά τους βασικούς τομείς. Μέσω ε, με την επιλογή αυτή έχετε τονίσει κάποια θέματα. Για παράδειγμα, βλέπουμε στις αεροδικέ μεταφορές ε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Όσον αφορά το σύνολο της ε, συζήτησης βρίσκουν ενδιαφέρον ότι τα κράτη-μέλη που έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση κατά 50% στους τομείς αυτούς, έχουν υποβάλει ένα σωρό ε, αιτήσει και εκπλήσονται όταν δεν γίνονται δεχτές οι αιτήσει τους. Ας ε, σκεφτούμε τι, πόσα χρήματα ήθελε το Κοινοβούλιο και πόσα τελικά ε, έλαβε. Πολλά προγράμματα λοιπόν δεν μπόρεσαν ε, να ληφθούν υπόψη. Πάντω βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα το αποτέλεσμα τη επιλογή. Αναφερθήκατε στο θέμα, στο πρόγραμμα ανάκαμψη. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι ιδιαίτερα λυπηρό. Θυμάμαι εποχέ κατά τι οποίε κάποιο πρόεδρο τη Επιτροπή, ένα κύριο Ζακ Ντελόρ, μιλούσε για τις ε, σημαντικές εργασίες ε, που προωθούν την Ευρώπη και θεωρούσε ότι τα έργα αυτά ήταν σημαντικά για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Εάν τώρα το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαψης για τις μεταφορές δεν λάβει ούτε ένα σέντς παραπάνω από τους πόρους που ήδη προβλέπονταν. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα στην Κομισιόν να συνειδητοποιήσουν ότι οι μεταφορές, η κινητικότητα και τα σχετικά προγράμματα πράγματι συμβάλλουν σε ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θετική ανάπτυξη και κατά 100% θα μπορούσαν να ταιριάξουν σε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης χωρίς να περιοριστούμε αποκλειστικά στους ε, πόρους ε, για τις μεταφορές. Και τέλος, ε, θα ήθελα να πω ότι για τα προγράμματα αυτά οι εξηγήσει που δώσατε ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Οι ερωτήσεις που έχω είναι ότι αναφερθήκατε στο ότι χρηματοδοτούνται εδώ 72% των προγραμμάτων που το 72% των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται είναι μελέτες. Τι γίνεται με τους πόρους που έχουν διατεθεί στο παρελθόν για μελέτες, από τις οποίες όμως δεν, προκέ... δεν προέκυψε εκ των υστέρων τίποτα. Τι έγινε δηλαδή με τα προγράμματα για τα οποία, στα οποία δεν δόθηκε καμία συνέχεια. Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε τα χρήματα αυτά. Ε, ο κύριος Αλκαντράουι. Ε, ε, ήθελα να συμφωνήσω με τον Ματιό. Αν δούμε τα επιλεχθέντα έργα, θα έλεγα ότι η επιλογή ήταν καλή. Δείχνουμε μια νέα τάση στον τομέα των μεταφορών. Ευνοούμε τους ιδιοδρόμους χρηματοδοτούμε με επιπλέον ποσά. Το RTMS επίσης χρηματοδοτείται πιο γενναιόδωρα, σημαντική μακρόπνοη κίνηση. Κάνουμε κάτι λοιπόν για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των μεταφορών μεταξύ άλλων. Όμως, όπως είπε και ο ανησυχώ για το μετά. Αποφασίσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος ανάκαμψης να επενδύσουμε ίσως λίγο πρόωρα προσδοκώντας όμως ότι στο τέλος της εφαρμογής αυτού του πολιετούς προεπολίσμου θα δούμε τι μένει και τώρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν μένει τίποτα. τώρα ερώτημα λοιπόν τι κάνουμε. Ποιες είναι οι πηγές επιπλέον χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων. Το να τα συνδυάσουμε, να φροντίσουμε να επικοινωνούν μεταξύ τους είναι σημαντικό. Είναι γνωστέ οι φιλοδοξίε των Ευρωπαίων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όμως τώρα το Ταμείο Μαργαρίτ, Μαργαρίτα, όπως το λέμε, δεν ξέρω και πολλά γι' αυτό μου λίγο καινούρια τα σχετικά. Όμως το ερώτημα είναι, θα μπορούσε το ταμείο αυτό, όπως έλεγα, προς το τέλος της περίοδου, επειδή θα έχουν αυτά τα ε, να χρηματοδοτήσει, να αντισταθμίσει την έλλειψη κονδυλίων. Μπορούμε εκεί να δεσμεύσουμε κονδύλια ακριβώς για τις μεταφορές. Thanks. Ευχαριστώ. Η κυρία Λιχανπέργερ κατευθείαν. Όχι, και θα επιστρέψω σε εσά, ε, κύριε Μάισνερ, μετά. Κυρία, κύριε Πρόεδρε, ήταν ενδιαφέρον το σχόλιο σχετικά με τα κονδύλια. Ε, φυσικά να συζητήσουμε και το που πηγαίνουν τα χρήματα αυτά εν μεταξύ. Τώρα, συζητούμε για τους αυτοκινητόδρομους, τις θάλασσες, Αυτό είναι το σλόγγαν, αλλά περί αυτού πρόκειται. Ξέρω ότι είμαστε εδώ για να μειώσουμε την γραφειοκρατία και φυσικά ξέρω ότι πρέπει να συγκεράσουμε και εθνικά συμφέροντα. Πολλέ χώρε περιμένουν αυτούς τους περίφημου αυτοκινητοδρόμου τη θάλασσα. εν πάση περιπτώσει, για να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά. Γιατί έχει καθυστερήσει η σχετική συζήτηση τόσα χρόνια, τη στιγμή που όλοι συμφωνούν. Φοβούμαι ότι δεν προχωρούμε παρά το γεγονό ότι υποβάλλονται προγράμματα, πολλά από αυτά όμω δεν είναι ρεαλιστικά. Λοιπόν, για να εστιάσουμε σε ρεαλιστικά έργα. Για να μπορέσουμε ακριβώ να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προ τα εμπρό. Έχω την εντύπωση ότι διάφορα κρατημέλη έχουν σκονισμένα στα συρτάρια του κάποια και κάθε φορά που περισσεύουν μερικά χρήματα λένε για να τα ρίξουμε στο τραπέζι. Και αυτό βλέπουμε έργα τα οποία έχουν απορριφθεί 3, 4, 5 φορέ. Ε, αυτά τα έργα δεν θα πρέπει να γίνονται καν αποδεκτά για συζήτηση. Η επόμενη Κομισιόν φοβούμαι ότι θα βρεθεί ε, μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων έργων. Λοιπόν, αν περισσέψουν υποδίλια, δεν υπάρχει κανένας λόγο να επανέλθουμε σε τέτοιου είδου ε, σκονισμένα έργα, να το πω έτσι. Και το λέω αυτό παρά το γεγονό ότι γνωρίζω ότι πίσω από μερικά από αυτά κρύβονται ισχυρά εθνικά συμφέροντα. Υπάρχει και το πρόσχημα ότι δεν πέρασε το έργο γιατί κάποιος άλλος έφταιγε. Τώρα, έχουμε μπροστά μας μια έκθεση για τα τέν. Είναι η έκθεσή μου που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Είχαμε αποφασίσει τότε να διαχωρίσουμε τους περιφερειακούς πόρους από τους άλλους για να έχουμε μια σαφή εικόνα των ποσών που ξοδεύονται εδώ. Γιατί πολλά έργα, ξέρετε, απορρίπτουν στο ένα ταμείο και μετά πηγαίνουν στο περιφερειακό ταμείο. Φοβούμαι ότι κάποιοι ψωνίζουν, όπως λέμε, επιλεκτικά ταμείο και κάθε φορά που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του ενός ταμείου τρέχουν για το άλλο. Αυτά τα πράγματα είναι παράλογα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι δεν παίρνουν τα καλύτερα έργα, αλλά τα έργα αυτών οι οποίοι ξέρουν, καλύτερα τα μέσα και τα έξω του συστήματος, των διαδικασιών. Τώρα, όσον αφορά τι εσωτερικέ θαλάσσιε, ε, εσωτερικέ υδάτινε οδού, υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ξέρω πολλά τέτοια έργα. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Υπάρχουν τέτοιου είδου περιπτώσει. Θα ήθελα να το ξέρω. Είναι πολύ... Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Έχω επίση την άποψη ότι μεγάλα κονδύλια πηγαίνουν σε δρόμου. Αλλά οι υποδομέ, οι οδικέ υποδομέ είναι πια τόσε πολλέ που αν αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτοκινητοδρόμους και δρόμους γενικότερα δεν θα τελειώσουν ποτέ. Τώρα για το Ταμείο Μαργκερίτ. Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια ποιος είναι ο στόχος αυτού του Ταμείου. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι είδους κερδοσκοπικές απόπειρες. Και εγώ θα κολλήσω αμέσω με το σχέδιο Μαργαρίτα, γιατί εγώ νόμιζα ότι αφορούσε μόνο στη Δανία. Υπάρχουν χιλιάδες μαργαρίτες στη Δανία. Λοιπόν, εμείς ε, το ξέρουμε ότι ως πολιτικοί των μεταφορών που είμαστε ζητούμε κάθε φορά ε, περισσότερα χρήματα. Ξέρουμε πολύ καλά τη σημασία των μεταφορών. Όλη η εσωτερική αγορά εξαρτάται από τις μεταφορές. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τους διαδρόμους. και είναι πολύ σωστή αυτή η επιλογή διότι μιλάμε πάντα και για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ε, μεταφοράς ε, και προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να δώσουμε αηφορία. Φυσικά είναι πάντα δύσκολο να γίνει η σωστή επιλογή. Ε, θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην πρόταση της κυρίας Πέρκερ. Ε, προτάσεις ε, που ε, επανειλημμένα υποβάλλονται και που έχουν πολύ ιδιαίτερο εθνικό χαρακτήρα να μην θεωρούνται παραδεκτές. Γενικά, θα μπορούσα να φανταστώ συγκεκριμένες προτάσεις να μην είναι τόσο επίγουσες, ωστόσο να είναι πολύ καλές. Και θα ήταν χρήσιμο να αποδεχτούν αυτές. Αυτό, αυτό το ξέρω την εμπειρία μου από το Κοινοβούλιο στην ε, Κάτω Σαξονία. Θα πρέπει νομίζω να γίνει διάκριση. Πρόκειται για τρελή πρόταση η οποία ε, έχει υποβληθεί ε, για, ε, για εθνικούς ε, για λόγους συμφερόντων ή είναι κάτι που γενικά ωφελεί την πολιτική μεταφορών. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ήδη υπόθηκαν πολλά από την ε, πολιτική μου ομάδα για το θέμα αυτό. Θα κλείσω λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ. Σύντομα, λέει ο κύριος Καντσάν. Σίγουρα εμείς ε, θα μιλήσουμε στην επόμενη περίοδο για το προγραμματισμό των ΤΕΝ. Αλλά Εμένα μου φαίνεται χρήσιμο, ξεκινώντας από το Ταμείο Μαργαρίτα, να μιλήσω για τον τρόπο χρηματοδότησης των υποδομών. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αντί να διαχέουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες θα πρέπει να τις συγκεντρώσουμε γύρω από τα διάφορα ταμεία, από τα διάφορα κονδύλια το Μαργαρίτα βρίσκεται υπό οικοδόμηση και θα ήταν πολύ χρήσιμο να χρηματοδοτούσαμε σημαντικά αυτό το ταμείο, διότι πέρα από το να ορθολογικοποιεί και να συμμετέχει στην υλοποίηση σχεδίων, ελέγχει και την κατασκευή τους Δηλαδή ότι για όλη την κατασκευή ακολουθείται διαφάνεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύστημα των ταμείων είναι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε έναν προγραμματισμό. Διότι εμείς θα πρέπει να έχουμε συνολικά ε, τον σχεδιασμό διότι πρέπει εμείς να ξεχωρίζουμε τον σχεδιασμό από το σύστημα κατασκευής. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ καλό σύστημα όπου έχουμε πραγματική συγχρηματοδότηση μέσα από το συνδυασμό ιδιωτικού και δημοσίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξανασυζητήσουμε το θέμα και στις επόμενες συνεδριάσεις που θα μιλήσουμε για το νέο προγραμματισμό αλλά θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει περισσότερο αυτό το, το, το, το μέσο και να κοιτάξει να υλοποιεί να, τα έργα κατά αυτόν τον τρόπο. Εμένα μου φαίνεται ότι στο Ταμείο Μαργαρίτα ε, συμμετέχει και το Ταμιευτήριο και το Ιταλικό ε, ταμιευτήριο και δεν αναφέρεται εδώ. Ε, νομίζω ότι όλα τα κράτη μπορούν, π, εκπροσωπούνται και δεν θα πρέπει να εκπροσωπούνται μόνο με δημόσιο χρήμα αλλά και με ιδιωτικά κονδύλια. Κυρία Γιάλα, εγώ θέλω να συγχαρώ καταρχήν την Κομισιόν διότι και πάλι μας, ε, έκανε, μας συνέταξε ένα σχέδιο πολύ δύσκολο Ε, το οποίο μας ε, οδηγεί, ε, μας βοηθά να προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Πακέτο εξής, έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένες προτάσεις που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε την αναθεώρηση των δικτύων, τη χρηματοδότησή τους και το μέλλον. Οπότε ρωτώ, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι όλα αυτά τα σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούμε και αν θα καταλήξουμε εμείς σε αυτούς τους στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει αυτή η λογική γραμμή μέσα στο πλαίσιο της οποία, που ακολουθώντας την προχωράμε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχουμε λίγα χρήματα, και οι μελέτες είναι αποτελεσματικές όταν πρέπει να κάνουμε μία αποτίμηση του κινδύνου. Ποιε, τι λένε οι μελέτες εδώ. Θυμούμε τον κανονισμό των δικτύων είχαμε προβλήματα με τον ορισμό των μελετών. Ε, θα ήθελαν η Κομισιόν να το εμβαθύνει κάπως περισσότερο για το πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι μελέτες για τη μείωση των κινδύνων. Για το Ταμείο Μαργαρίτα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καντσάν. Είναι πολύ καλό που καταφέραμε να συμμετέχουν οι μεταφορές Θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Σίμψον αν κάποια στιγμή σε αυτήν την επιτροπή που μπορεί εγώ να το χάσα βέβαια μπορεί ήδη να έχει γίνει αλλά τέλος πάντων πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μία παρουσίαση, αναλυτική παρουσίαση αυτού του ταμείου και το πώς συνδέεται με όλες τις πλευρές της κινητικότητας, της συνοχής, της ασφάλειας στις μεταφορές. Λοιπόν, το ψάχνα εγώ το σχέδιο Μαργαρίτα να πάρω πληροφορίες και μου ήρθε έτσι μπροστά μου τώρα. Και για το σχέδιο Easy Way που παρουσιάζει η Κομισιόν. Μας δίνετε τον προγραμματισμό που είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια των ITS, αλλά θέλω να ξέρω τι γίνεται για τη φάση 1. Μπορείτε να μας δώσετε διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα ο κύριος Λιμπεράτσικη. Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω τρεις προτεραιότητες, οι οποίες είναι σωστά επιλεγμένες. Άκουσα αυτές, όμως έχω ένα ερώτημα στη σελίδα 6 παρουσιάζετε τις προτεραιότητες και τα ποσά και λέτε ότι έχουμε 370 εκατομμύρια τα οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί ως τα 357 μας μένουν 13 λοιπόν ακόμη Αυτά θα τα δώσουμε ή δεν υπάρχουν ακόμη, δεν υπάρχουν άλλα επιλέξιμα έργα για χρηματοδότηση. Για να δούμε εδώ πώς έχει το πράγμα. Τώρα, σύμφωνα με τις αιτήσει που λάβαμε, βλέπω 12 τελικά 12 ισπανικά έργα. Η Πολωνία έχει υποβάλει μόνο τρία έργα, αν και παρομοίου μεγέθους, όσον αφορά την έκτασή της τουλάχιστον με την Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχε ε, αιτήσει, αντίστοιχε με τι ανάγκε. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, πώς το σχολιάζετε. Συγχαίρω βεβαίω την Ιταλία γιατί υπέβαλε έργα αξίας 69 εκατομμυρίων. Στην Πολωνία ήμασταν στα 6,3 μόνο εκατομμύρια. Το επόμενο ερώτημά μου είναι τι κάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τι αιτήσει, εξωτερικοί ανεξάρτητοι πυρογνωμόνε αξιολογούν τι προτάσει και στη συνέχεια η Κομισιόν εγκρίνει την γνωμοδότηση των ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων και δημοσιεύεται αποτελέσματα. Εμπλέκεται επαρκώ η Κομισιόν, ασχολείται με το θέμα. Ευχαριστώ. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să um, atrag atenția asupra câtor... Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια βασικά στοιχεία. Καταρχήν, για το ετήσιο πρόγραμμα 2009 και στα πλαίσια του πολιετούς προγράμματος έχουν ε, δοθεί πολλοί πόροι, έχουν διατεθεί πολλοί πόροι και ένα μέρος αυτών διατίθεται για τις ε, εγγυήσεις ε, των πιστωτών. 5,7 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ζητήθηκαν. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τα, 2000, για τα έτη 2010 με 2013 ένα δισεκατομμύριο θα μείνει μόνο για τα προγράμματα TNT. Αυτό σημαίνει 240 εκατομμύρια το χρόνο. Αν εξετάσουμε τα σχέδια ε, για τις ε, υποδομές θα διαπιστώσουμε ότι αυτό είναι σχεδόν τίποτα. Να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν, τι θα κάνει στον τομέα των μεταφορών με τον προϋπολογισμό αυτό. Μία πρόταση για τον Πρόεδρο. Θα ήταν ενδιαφέρον η Επιτροπή μας Μεταφορών και Τουρισμού την επόμενη χρονιά, το πρώτο εξάμεινο ενδεχομένω, να οργανώσει διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να συζητήσουμε την χρήση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στην επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών και ενδεχομένω να διαθέσουν περισσότερου πόρου ε, για έργα υποδομή. Ε, και επίση ε, ω προ τη διαδικασία επιλογή. Θα ήθελα να ζητήσω το εξή από την Κομισιόν. Θα ήταν χρήσιμο και τα κράτη-μέλη να ακούσουν. Πρόκειται για την πρόσβαση στην ιστοθέση TNT. Θα ήταν χρήσιμο εάν αναφέρονται εκεί τα προγράμματα που επιλέχθηκαν. Και αναφέρομαι εδώ στο περιεχόμενο των αιτήσεων, διότι είμαι πεπισμένη ότι και άλλα κράτη-μέλη που μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να επιλεγούν τα, προγράμματα, τα προγράμματά τους, να αποκτήσουν μια εικόνα σχετικά με το ποια προγράμματα έχουν επιλεγεί τα προηγούμενα χρόνια. Επανέρχομαι στις δύο αποφάσεις για το πολιετές πρόγραμμα και το ε, ετήσιο πρόγραμμα. Να ε, αναφέρω την περίπτωση της Ρουμανίας έχω διαπιστώσει από το, για το 2009 η Ρουμανία δεν έχει υποβάλει καμία αίτηση για το πολιετές πρόγραμμα. Η Ρουμανία ε, πρότεινε προγράμματα μεταξύ άλλων ένα που συνδεόταν με το Motorways on the Sea για την Μαύρη Θάλασσα. Ίσως ε, να είναι κάπως ε, περίεργη η παρουσίαση, διότι αναφέρεται ότι επειδή δεν υπάρχουν ε, άλλα έργα από την ε, περιοχή αυτή, το οποίο ουσιαστικά θα σήμαινε προστιθέμενη αξία, για το λόγο αυτό απορρίφθηκε το πρόγραμμα, επειδή δεν υπήρχαν άλλα προγράμματα από την περιοχή αυτή. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν καθόλου ε, προγράμματα για την Μαύρη Θάλασσα. Αυτό βρίσκω ότι είναι λάθος, διότι για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία η Μαύρη Θάλασσα είναι πολύ σημαντική περιφέρεια και γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο από την αρχή να ε, συμμετέχουμε και να γίνει αποδεκτό ένα πρόγραμμα από την ε, περιοχή αυτή για να πετύχουμε προστιθέμενη αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Μαύρη Θάλασσα λοιπόν. Και γι' αυτό μου φαίνεται περίεργη η απόφαση αυτή όσον αφορά το Ταμείο Μαργκερίτ. Και θα κλείσω τις παρατηρήσεις μου. Το ταμείο αυτό ε, δημιουργήθηκε ε, στα πλαίσια της καταπολέμησης της αλλαγής του ε, κλίματος για να κατανεμηθεί η προσπάθεια. Πρόκειται για πόρους, για οικολογικές μεταφορές, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Τικάου. Και τέλος, εγώ θα ήθελα να πω ότι προσπάθησα να διαβάσω τα δύο αυτά κείμενα και να βρω χρήσιμα έργα τα οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν την Βόρεια με την Νότια Ιρλανδία. Τα διάβασα τέσσερις φορές και δεν βρήκα ούτε ένα. Κατανοώ γιατί ο κ. Σιμπεράτσκι αισθάνεται απογοητευμένος με τα τρία, αλλά είναι τρία πάνω από το μηδέν το 0 του Ηνωμένου Βασιλείου. Σωστά είπε και η Μαύρη Θάλασσα κυρία Τικάο και δεν ξέρω αν φταίει τώρα η Ρουμανία ή ποιος άλλος αλλά εμείς υποβάλαμε αιτήσεις και δεν πήραμε τίποτα. Το 902.1 ο τοπικός σιδηρόδρομος που θα έλυνε τα προβλήματα στο Μάντσεστερ δεν εγκρίθηκε. Οι Γερμανοί λένε πολύ απλά τη λέξη στα γερμανικά απίστευτο. Απίστευτο που απορρίφθηκε αυτό το έργο. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους πραγματικά. Καταλαβαίνω γιατί οι Ισπανοί και οι Ιταλοί τα πήγαν τόσο καλά. Και φαντάζομαι, καταλαβαίνετε και εσείς γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω την κατάσταση εδώ. Φυσικά, καμία απόφαση δεν είναι τέλεια, αλλά τι να σας πω, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με τις αποφάσεις. κ. Λιμπεράτσκι ρώτησε, τι γίνεται, τα δίνετε στους εμπειρογνώμονες, αξιολογούν και συγκρίνετε. Όχι, αλίμονο. Ε, Οι εμπειρογνώμονες είπαν ότι το 1921, μεταξύ άλλων θα πρέπει να έχει εγκριθεί, αλλά ε, μας λένε ουσιαστικά ελάτε σε πέντε χρόνια, να τα ξαναπούμε, όταν θα έχουμε χρήματα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, δυστυχώ. Γι' αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι οι ορισμένα κρατημέλη δεν πήραν τίποτα και η χώρα μου είναι μία από αυτέ. Γιατί αν δεν κάνω λάθος η Βόρεια είναι τμήμα του Ινωμένου Βασιλείου, είναι σε άμεση επαφή με την Νότια αλλά ούτε και αυτή πήρε τίποτα. Θα είμαι ειλικρινή για μια σα. Η απόφαση του 1902-1 ήταν μια γελία απόφαση. Λοιπόν, επόμενο τέρμα οι διπλωματικέ εκφράσει. Πρόεδρε, θα παρήσω στις ερωτήσεις μία προσμία. όπως και να τις πάρετε, να φροντίσετε να έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μου, μέχρι τις 5.30. Πρόεδρε, θα απαντήσω σε όλες και θα είμαι και σύντομος για να καλύψω ακριβώς τα πάντα και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεχνούσα να απαντήσω στη δική σας ερώτηση. Οι βουλευτές ανέφεραν το follow-up των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν με συγχωρείτε. Ορισμένοι σχολίασαν το υψηλό ποσο των μελετών. Θα ήταν χρήσιμο αν σα δίναμε έναν ξεχωριστό κατάλογο που χρηματοδοτήσαμε την περιοδο 2002 2000-2006 για να δείτε και το αντίστοιχο follow-up. Δεν έχω τι στατιστικέ αυτές αυτή τη στιγμή, πρόχειρες. είτε ότι θα τις δούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάντως από κανονιστική απόψεω δεν υπάρχει επίσημη υποχρέωση για ένα μέλο, μέλος από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια μελέτη να συνεχίσει με έργο. Κοιτάξτε, οι μελέτε δεν είναι απλώ χαρτιά. Πρόκειται για μελέτες οι οποίε είναι προπαρασκευαστικέ μελέτες που αφορούν τη σύραγγα λιόν το Ρήνο, την Μπρένερ και το καθεξής. Είναι μελέτες που ακολουθούν άλλες που έχουν κοστίσει πολλά εκατομμύρια και θα υποστήριξουν από εδώ και πέρα τη δημιουργία της α, η οποία θα γίνει προπαρασκευαστικά εν ώψη της κατασκευής του κυρίου έργου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μελέτες οι έχουν και υλικό περιεχόμενο και οι οποίες προηγούνται του κυρίου κατασκευαστικού έργου. Πάντως είναι χρήσιμη προτασή σας θα συντάξω ένα συγκεντρωτικό κατάλογο και θα τον στείλω στην Επιτροπή σας. Και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος του προγράμματος, το ανέφεραν και αυτό πολλοί βουλευτές, τα υπολοιπόμενα κονδύλια είναι πολύ λίγα, λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο, ακόμα και αν τα βάλει όλα μαζί. αν και στην πραγματικότητα είναι ακόμα λιγότερα, γιατί έχουμε προκαταβολές 500 περίπου εκατομμύρια να πληρώσουμε. Αν δείτε τώρα τα 5 δισεκατομμύρια του 2010 που είχαμε προκρίνει το 2007 μαζί με το Κοινοβούλιο, αυτά θα αναθερθούν του χρόνου. Από αυτά ελπίζουμε ότι ένα μικρό ποσοστό θα κρατεί διαθέσιμο γιατί κάποια έργα δεν ξεκίνησαν, άλλα δεν ολοκληρώθηκαν κλπ. Άρα θα προκύψει ένα διαθέσιμο ποσό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι διαχειριζόμαστε τα κονδύλια αυτά με τρόπο ικανοποιητικό όπως κάνουμε κάθε χρόνο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και εν πάση περιπτώσει όταν κάτι δεν χρησιμοποιείται θα το πηγαίνουμε αλλού το χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς άλλου έργου. Ελπίζω λοιπόν πολύ σύντομα ότι θα μπορέσω να υποβάλω σε εσά μια επισκόπηση του τι μένει γενέστε μέχρι το του προγράμματος και θα σας καταθέσω και τις προτεραιότητες για την περίοδο 2011-2013 όσον αφορά τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, εδώ δεν έχουμε τρέξει όσο μπορούσαμε. Κρίμα, αναζητούμε τις αιτίες για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα κρατημέλη και να υποβάλουν και αυτά με τη σειρά τους καλύτερα έργα. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει και την εργασία της για την ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων, των θαλασσίων αυτοκινητοδρόμων. Συνεχίζουμε να προβλέπουμε, να διαγωνισμοποιήσει τα έξυπνα μεταφορών. Δεν ξέρω πώ θα προχωρήσει αυτό. Θα χρειαστεί μία εκ των υστέρων αξιολόγηση του Easy Way, της φάσης 1. Και βάσει αυτή τη αξιολόγηση θα προετοιμάσουμε την απόφαση χρηματοδότηση της φάσης 2 με βάση την απόφαση επιλογής. Η απόφαση επιλογής βεβαίως αφορά ένα ανώτατο όριο, δεν είναι η, απόφαση, η τελική απόφαση που θα λάβει η εκτελεστική επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο, όπως έγινε για την φάση 1. Έχουμε λοιπόν τις εγγύσεις, έχουμε του θαλασσιούς αυτοκινοδρόμους. Έχουμε ένα κομμάτι που αφορά πληροφορική και τηλεπικοινωνίες και θα δούμε τι θα μείνει για τα τακτικά ετήσια προγράμματα. Ούτως ή που πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο ανεξαρτήτως του πόσο λίγοι είναι διαθέσιμοι πόροι, είναι ένα πρόγραμμα ελκυστικό θα χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό και θα τον εξαντλήσουμε. Τις μελέτες θα συνεχίσουμε να τις χρηματοδοτούμε. Το ποσοστό χρηματοδότηση είναι 50%. Το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από τα κρατημέλη. Έχουμε κατά τα άλλα καταστρώσει και τα προγράμματα έως και για το 2013. Αυτά φυσικά δεν είναι αρκετά. Συμφωνώ. Όπως είπατε πρέπει να κάνουμε επιλογές δύσκολες. Θεωρώ όμως ότι έχουμε καταδείξει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Εκεί που καθυστερούμε είναι ότι οι κρατικοί, οι εθνικοί πόροι δεν τρέχουν παράλληλα με τις αιτήσει τους. Φυσικά στις επόμενες ε, χρηματοοικονομικές προοπτικές θα ξανασυζητήσουμε το θέμα. στο. το πρόγραμμα προχωράει με βάση τους στόχους οι οποίοι προκρίθηκαν με διαφάνεια. Πέρα από την γενικότερη πολιτική φυσικά υπάρχουν και ενδιάμεση στόχοι, ενδιάμεσα στάδια, με φορμή τα οποία θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ενδεχομένως και υψηλότερη χρηματοδότηση. Τώρα, θα θέλαμε έναν τρίτο διαγωνισμό ERTMS. Δεν είναι βέβαιο αυτό. Στις προηγούμενες φάσεις νομίζω πήγαμε καλά. Και αυτό θα μας επιτρέψει να περάσουμε και στην περίοδο 2018 έως 20. Τώρα άκουσα σχόλια για το Μαργκερίτ. Κοιτάξτε, είναι το ταμείο το οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και διάφορα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες μέλη. Η Ιταλία υποστηρίζει την προσπάθεια με το ταμιευτηριό της δεν έχω πιο πολλά να σας πω γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος. Πάντως ο διαγωνισμός, ο σχετικός διαγωνισμός είναι ακόμη ανοιχτός. Και εκτιμάται σαφώς ότι διάφοροι οργανισμοί από διάφορες χώρες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Μαργκερίτ. Ο βασικός στόχος είναι να μαζέψουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να έχουμε μια δεξαμενή κονδυλίων για να χρησιμοποιήσουμε έρευνα, διευρωπαϊκά δίκτυα, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, υποδομέ και ούτω καθεξής. Το ταμείο αυτό θα ασχολείται κατά κύριο λόγο με έργα τα οποία θα προάγουν την υψηλή απόδοση έργων, έργων για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Δεν υποκαθιστά το Ταμείο τις άλλες χρηματοδοτήσεις, όμως βάσει τη συμφωνία μεταξύ Ταμείου και Κομισιόν, τουλάχιστον 80 εκατομμύρια θα πάνε σε διευρωπαϊκά δίκτυα. Έρχονται και επιπλέον κονδύλια, δεν ξέρω πόσα. Πάντω να έχετε υπόψη σα ότι επειδή τα, η σχέση χρηματοδότηση δανείων είναι προ 5, εμεί χρηματοδοτούμε μόνο το 15% περίπου, οπότε μπορείτε να φανταστείτε το συνολικό ύψος των επενδύσεων για όλα αυτά τα έργα. Έργα εξαιρετικά διαφορετικά. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν είναι βεβαίως υποκατάστατο των πάντων, έτσι. Τώρα, αν βάσει της πολιτικής των ταμείων και των τεν ε, ψάχνουμε όλοι να χρηματοδοτήσουμε έργα ανεξάρτητα το αν κολλάνε ή δεν κολλάνε. Κοιτάξτε, είναι θέμα επιλεξιμότητας. Για τις μελέτες πολλοί έρχονται στα τέν των μεταφορών και για τα έργα πηγαίνουν σε άλλα ταμεία. Άρα δεν πρόκειται για κατάχρηση, καταχρηστική επιλεκτική συμπεριφορά, αν θέλετε. Και να απαντήσω σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, να αρχίσω να απαντώ. Το ότι κάτι δεν είναι ότι δεν είναι καλό έργο. Υπάρχει υψηλός σκληρός ανταγωνισμός και υπάρχουν χρηματοδοτικοί περιορισμοί. Φυσικά από αυτά που είναι κάποια δεν είναι αρκετά ποιοτικά αν θέλετε, από τους ανεξαρτητούς εμπειρογνώμονες ή εν τέλει δεν προκρίνονται από την ε, Κομισιόν βάσει των κριτηρίων και των προτεραιοτήτων που σας ανέφερε. δηλαδή τον περιορισμένο προπολογισμό καταρχήν όπως έγινε και με το Manchester δυστυχώ. Αυτό απαντά και στην ερώτηση περί εξωτερικών ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων. Φέτος, κοιτάξτε, οι εμπειρογνωμόνες έκαναν την προπαρασκευαστική δουλειά, βαθμολογούν μαζί με το εκτελεστικό όργανο του ΤΕΝΤΗ τα έργα για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά από τη στιγμή που έχουν κάνει την πρώτη εξέταση και έχουν αξιολογήσει το έργο βάσει των γνωστών κριτηρίων. Το παιχνίδι πιάνει στα δικά μα χέρια και εκεί πρέπει να κάνουμε δύσκολε επιλογές, να πάρουμε δύσκολε αποφάσεις. Και τα αποτελέσματα και τα περίπτωση ικανοποιούν ή δεν ικανοποιούν κάποιους. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν, δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα το εύκολο να καλύψουμε ομοιόμορφα όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό τα λέμε κάθε χρόνο, αυτά ισχύουν σήμερα και θα ισχύουν και αύριο. Πάντως τα έργα που επιλέξαμε είναι καλά έργα και να ξέρετε ότι δεν θα είχαν επιλεγεί αν δεν ήταν τόσο καλά. Τώρα για, το, τα έργα που υποβάλλονται μία, δύο, τρεις, πέντε φορές δεν προβλέπεται σχετικά από τον κανονισμό και ξέρετε είναι πιο εύκολο να επανυποβληθεί ένας φάκελος είναι κατανοητό αυτό έχω και στο μυαλό μου αυτό το οποίο υπονήσετε και εσείς αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά δεν έγινε αυτό που έγινε δηλαδή για να παρακαμφθούν οι κανόνες εν πάση περιπτώσει θέλω ξανακοιτάξω όμως το ζήτημα και τώρα να ρίξω μια ματιά εδώ, μήπως ξέχασα κάτι. Για το Μαργκρίτ νομίζω τα είπαμε. Αν θέλετε φυσικά, αν θέλει η Επιτροπή σας, η Κομισιόν είναι εδώ να σας πει περισσότερα. Μπορούμε να ξαναρθούμε την γενική μου διεύθυνση και θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να συζητήσουμε όλοι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι πατέρας του Μαργκερίτα, αν θέλετε. Και τώρα θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι, όπου θα παρουσιάσα και εγώ την κατάσταση, εξέφρασα τη λύπη που προχωρήσαμε. Μας λείπουν όντω μετά τα 570 τα υπόλοιπα 13 ε, εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται τμήμα του προπολογισμού. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά ούτως ή άλλως. Οι αποφάσει ένταξης είναι αποφάσεις πλαίσια με βάση τις οποίες κινείται και το Ταμείο κάθε χρόνο. Ο σκοπός είναι να μην χάνονται χρήματα και δεν χάνονται. Τα χρήματα αυτά που δεν εξοδεύτηκαν το 2009 θα παραμείνουν στον κορβανά μας το 2010 όχι άσχημο δεδομένη και της έλλειψης κονδυλίων που θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί έγινε. Θέλησαμε να περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά περισσεύει κάποιο ποσό. Τώρα για τους αυτοκινητοδρόμους. είναι προτεραιότητα, το ξέρετε αυτό. Και είναι κρίμα που μια σχετική μελέτη δεν εγκρίθηκε. Δεν θυμάμαι αν έγινε αυτό επειδή το απέρριψαν ε, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονε ή επειδή η Κομισιόν το απέρριψε στην ε, συνέχεια. Η ξεκίνησε από θερική γνωμοδότηση και μετά απορρίφθηκε. Ε, Ξέρετε, ένα έργο το οποίο υπορρίφθηκε η αιτιολογία υπάρχει στι εξηγήσει της σχετική απόφαση. Αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο δείτε για ποιο λόγο ακριβώς και πώς απορρίφθηκε η συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί ήταν ένα χρήσιμο, σαφώ ένα καλό έργο, απλώ δεν ήταν αρκετά όριμο. Πάντω, εμεί στέλνουμε συστηματικά στα κράτη-μέλη, στις αξιολογήσεις όλων των έργων για να ξέρουν γιατί εγκρίθηκαν, γιατί απορρίφθηκαν, γιατί κάποια καλά σχέδια δεν εντάχθηκαν τελικά. Βάρος παρακολουθούμε τα, την ποιότητα των έργων, η οποία βελτιώνεται από χρόνο σε χρόνο. Πρέπει μάλιστα να σας πω ότι φέτος είχαμε περισσότερες αιτήσεις από ποτέ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε όλοι και βελτιώνεται και η παρουσίαση των αιτήσεων. Τώρα για το Ενωμένο Βασίλειο. έγκριναμε καταρχήν ένα ναι στην Ολλανδία και παρουσιάμε άλλα τρία ή τέσσερα. Όπως είπατε, τώρα που ξεκίνησε και το Ενωμένο Βασίλειο να υποβάλει προτάσεις, θα προχωρήσει. Στα 500 εκατομμύρια του Ιουλίου, μάλιστα, το πήγε ιδιαίτερα καλά το Ρωμανικό Βασίλειο. Δεν έχω εδώ τι λεπτομέρειε, δεν έχω το προσπέκτου, αλλά νομίζω ότι πήραν περισσότερα από ό,τι σε όλη την ιστορία των χρηματοδοτήσεων στον τομέα αυτών. Τα ποσά ήταν αρκετά, μην νομίζετε. Μιλώ για αρκετά υψηλά ποσά. Και τώρα, συγκεκριμένα, για τα συγκεκριμένα έργα, ο κόμβος στο Μάντσεστερ. Θεωρήσαμε ότι η, στάση, η μελέτη θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αλλά υποβλήθηκε καθυστερημένα. Και το κυριότερο ήταν το θέμα της δανειοδότησης 560 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε μια μεγάλη διαφορά και ξέρετε, όταν έρχεται η ώρα να παίρνει κανείς αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις, θέλουμε να προκρίνουμε προτάσεις που έχουν εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τα δάνεια. Δεν πιστήκαμε λοιπόν προκειμένου εδώ. Στήριζονταν υπερβολικά το έργο σε κοινωτικά χρήματα. Πρώτα το μόνο που έχω να πω στο σημείο αυτό είναι ότι κάποια έργα εγκρίθηκαν από τα 250 εκατομμύρια τα, 80. Ε, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, υπάρχει ανταγωνισμό και προκρίνουμε τα έργα τα οποία είναι καλύτερα, θέλετε, πιο ενδιαφέρονται σε σχέση με άλλα. Κύριε να σα ευχαριστήσω, αν και δεν πείθαμε από όλα σα τα επιχειρήματα. Σα ευχαριστώ για την απάντησή σα. 658.000 ζήτησαν, όχι 658 εκατομμύρια. Επασεπτό, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα στην συνεδρίαση των συντονιστών. Ναι,